Borrell isn't in yet. Yes. Oh, he's, oh sorry, I haven't seen him. Okay, okay. Dear colleagues, good morning. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε παρακαλώ να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Directly to point three, I will make later the announcement. Πάμε στο 3, αφήνω τις ανακοινώσεις για αργότερα πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίε για την καταπολέμηση τη νομοποίηση εισόδων από παράνομε δραστηριότητες. Εξέταση των τροπολογιών. Η συγκητή μα είναι ο Εμμανουέλ Μορέλ. Κατατέθηκαν 52 τροπολογίε. και ο εισηγητή θα καταθέσει τρει συμβιβαστικέ τροπολογίε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Μορέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κινητοποιηθήκαμε ιδιαίτερα για την φορολογική δικαιοσύνη. Είχαμε τι δύο επιτροπέ ΤΑΞ, την Επιτροπή για τα έγγραφα του Παναμά και κάποιε ενδιαφέρουσε προτάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι που δείχνει ότι όταν ασκείται πίεση από την κοινή γνώμη και μια κινητοποίηση των Ευρωβουλευτών, τα κοινοτικά θεσμικά όργανα αφουγκράζονται αυτές τις ανησυχίες και σε αυτή την ε, σχετικά ζωφερή και θλιβερή περίοδο είναι θετικό ότι αν άλλο αυτό το θέμα προχωρούμε. Στο θέμα της φορολογικής διαφάνειας ε, έχουμε από τα πιο σημαντικά και ζωτική σημασία ε, θέματα, γιατί ο κόσμος έχει εξοργιστεί από τις αδικίες ε, που όλο και εντείνονται και δημιουργούν μια εύλογη δυσαρέσκεια. Και μάλιστα βασικές αρχές της δημοκρατίας είναι η ισότητα απέναντι στον νόμο και στη φορολογία. Γι' αυτό χρειάζονται κάποιε αλλαγέ, αυτέ που προτείνουμε και που θα ενταχθούν σε μια σειρά οδηγιών που βαίνουν προ τη σωστή κατεύθυνση. Διαπιστώνω με χαρά ότι συμφωνούμε όλοι για την ε, ε, ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για την νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε και τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία και ευχαριστώ του και ηγητέ των διαφόρων ομάδων για τη συνεργασία του. Θέλουμε εξασφάλιση των πληροφοριών στις, ε, των εφοριών κάθε κράτου και επίσης ε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το φορολογικό σχεδιασμό και αυτό και θέλουμε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Το κείμενο με τις τροποποίησεις ε, είναι ισορροπημένο, χάρη και στην συμβολή των σκιωδών εισηγητών και έτσι καταφέραμε ε, να εμπλακούμε στις διερευνητικές αυτές αποστολές. Θέλουμε να δείξουμε ρεαλισμό γιατί η αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων προϋποθέτει μία προετοιμασία των φορολογικών διοικήσεων και άρα σωστό εξοπλισμό τους. Και μέχρι τον επόμενο χειμώνα έχουμε την ευκαιρία για να θεσπίσουμε την νέα αυτή οδηγία. Και να τη βάλουμε στα σκαριά. Νομίζω ότι ε, υπάρχει όλο και αυξανόμενη απέτηση για φορολογική δικαιοσύνη και ανταποκρίνεται και η πρότασή μας σε αυτό το εύλογο αίτημα. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βαντέγκεντερνάρ, τον σκιώδη του ΕΛΚ. Ευχαριστώ και καλημέρα συνάδελφοι. Θα είμαι σύντομος και αποτελεσματικός. Όπως και η διαδικασία άλλωστε ήταν σύντομη και αποτελεσματική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ γρήγορη δουλειά που έκανε. Συμφωνούμε πράγματι ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ μικρή αλλά ουσιαστική αλλαγή στην νομοθεσία για να καταπολεμήσουμε τη νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε, οπότε θα πρέπει να επικεντρωθούμε στου ελέγχου και στη συλλογή πληροφοριών και με συνέργειες οι οποίες θα πρέπει πραγματικά να τι εκμεταλλευτούμε πλήρως. Εδώ πέρα λοιπόν δίνουμε προτεραιότητα στην γρήγορη υιοθέτηση της ε, πρότασης της Κομισιόν. Γι' αυτό ακριβώς ε, θα υποβάλουμε και κάποιες τροπολογίες για να υποστηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν. Επίσης, ε, συμφωνούμε ότι οι πληροφορίες για τον πραγματικό ιδιοκτήτη πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλες τις αρμόδιες αρχές. Και αυτό η ομάδα μου θα στηρίξει ένα κείμενο για να μοιραστεί η πληροφορία αυτή αυτομάτως μέσω του συστήματος αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Από το ECR. Η κυρία Προχώνερ Λέρνερ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή μας τον κύριο Μορέλ για τις πολύ καρποφόρες διαπραγματεύσεις και τις πολύ ισορροπημένες συμβαστικές τροπολογίες. Κατά τη γνώμη μου τώρα δημιουργούμε ένα πραγματικό πλαίσιο για διαφανή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων. Αυτό είναι και το ζητούμενο άλλωστε. Και ελπίζω οι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσουν αυτή τη διαφάνεια, τη φορολογική και την συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Το ένα από τα προβληματικά θέματα ήταν η πρόσβαση των εφοριών σε πληροφορίε για την καταπολέμηση τη νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Θα πρέπει να εναρμονιστούν αυτέ οι πρακτικέ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ με τι τροπολογίε μου θα δώσω έμφαση στο καθήκον που έχουν διάφορε δικαιοδοσίε να διερευνούν πληροφορίε που λαμβάνουν το συντομότερο δυνατό ασχετά με την πηγή αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, θα ήθελα τα κράτη-μέλη να έχουν την υποχρέωση να κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν μπορούν για τον ΑΒ λόγο να διεξαγάγουν έρευνες με βάση τις πληροφορίες που έλαβαν. Έτσι αποτρέπονται οι φορολογικές διοικήσεις ε, από τον πειρασμό να θελοτυφλήσουν ε, όταν λαμβάνουν κάποιες πληροφορίες. Επίση, τέτοιε πληροφορίε για την ε, νομοποίηση εισόδων από παράνομε δραστηριότητε θα πρέπει να εμπίπτουν στην υποχρέωση, στην υποχρεωτική ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Ευχαριστώ, κύριε Στόρβαλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε τον εισηγητή. Νομίζω ότι καταφέραμε να βελτιώσουμε κάπως τα πράγματα. Ταυτόχρονα όμως φοβάμαι ότι αφήνουμε πολλά παραθυράκια. Τέτοιου είδου νομοθεσία έπρεπε να υπάρχει ήδη από το 2003. Όταν τέθηκε σε ισχύ η οδηγία για τις τράπεζες, επειδή αυτή η οδηγία για τις τράπεζες ουσιαστικά οδήγησε στην ε, έξοδο ανθρώπων ε, γεγονός που δείξε στα Panama Papers. Αν δείτε την Task Force ε, για τη χρηματοπιστωτική δράση και τι κάνουν και την τοποθεσία σελίδα έχουν καταφέρει να εντοπίσουν ε, τη Βόρεια Κορέα που δεν είναι το κεντρικό κομμάτι του προβλήματος. Αν δείτε τα καζίνο, πιστεύω ότι τουλάχιστον το 60% του κύκλου εργασιών ε, των καζίνο προέρχεται από άγνωστες πηγές. Και ένας λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτό το παραθυράκι είναι ότι ουσιαστικά το δικαίωμα της λήθης ε, αφαρμόζεται στην περίπτωση των καζίνο. Έχουμε λοιπόν νομοθεσία που ουσιαστικά ε, φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Επίσης γνωρίζουμε ότι η διαδικασία της δέωσας επιμέλειας δεν ανταποκρίνεται στα απαραίτητα πρότυπα. Απλά στην προκειμένη περίπτωση βελτιώνουμε λίγο τα πράγματα και ελπίζω να συνεχίσουμε προς την ίδια οδό και για το μέλλον, διότι θα χρειαστούμε πολύ σκληρότερα εργαλεία ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε όλα τα παραθυράκια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Διάγκας. Όχι. Μαλή Σκότ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Μανουέλ για τι εξαιρετικέ του προσπάθειε. Η προτινόμενη νομοθεσία, όπω είπε, είναι κρίσιμη σημασία για την παροχή πληροφοριών στι φορολογικέ αρχέ για την καταπολέμηση της ε, φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Θα πρέπει να επισημάνουμε ζητήματα που μπορούν να βελτιώσουν την νομοθεσία και το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι φορολογικέ αρχέ. Συνεπώ, υποστηρίζουμε δύο από τα κύρια ζητήματα που υπάρχουν στι συμβιβαστικέ τροπολογίες του εισηγητή. Πρώτα απ' όλα είμαστε υπέρ τη αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση με την οδηγία νομοποίησης εσόδων παρόμοιε δραστηριότητε μεταξύ φορολογικών αρχών, γεγονό που θα ωφελήσει στην καταπολέμηση των διασυνεριακών ε, περιπτώσεων ε, απάτη και επίση θέλουμε η Κομισιόν να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Επίσης θα ήθελα να αφιερώσουμε λίγο χρόνο και στις δικέ μας ε, τροπολογίες που θεωρούμε ότι μπορεί να υποστηριχθούν και από άλλες ομάδες στις 35 και 42 προτείνουμε να δίδεται στις φορολογικές αρχές η δυνατότητα ερευνών εγχώρια με σκοπό την απόκτηση επιπλέον πληροφοριών όταν ένας φορολογούμενος της ε, τούσες αρχής ε, εμπλέκεται. Αυτό υπάρχει ήδη στην οδηγία για τη διοικητική συνεργασία. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα ήταν πολύ αποτελεσματικό τέτοιου είδους φορολογική συνεργασία πράγματι να λαμβάνει χώρα και μεταξύ φορολογικών αρχών. Στην τροπολογία 49 προτείνουμε διεύρυνση του αντικειμένου των στοιχείων ε, στα οποία μπορούν να έχουν προσβάσει φορολογικές αρχές. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες ε, που περιλαμβάνονται από την οδηγία EMLD όπως εξολογής κινδύνου, πληροφορίες δέωσης επιμέλειας των πελατών. Αυτό μπορεί να ωφελήσει ε, στην ανείχνευση της φοροδιαφυγής. Επίσης σας καλούμε να υποστηρίξετε την τροπολογία 15 που συντάξαμε βάσει απόψεων εμπειρογνωμόνων για να βοηθήσουμε στην επίτευξη ε, του στόχου αυτής της οδηγίας. Η τροπολογία αναφέρει διάφορα παραθυράκια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την παράκαμψη της ε, αυτόματης ανταλλαγής στοιχείων και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή ε, αυτής της έκθεσης ώστε να επισημάνουμε τα ζητήματα αυτά, ώστε να ξεκινήσει μια συζήτηση για να αντιμετωπίσουμε τις πιθανές αδυναμίες της ε, τρέχουσας οδηγίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μάρκο Τζάνι δεν είναι εδώ. Ο κ. Ευχαριστώ. Και εγώ προσυπογράφω τη συμφωνία που μας παρουσιάζει ο κύριος Μορέλ. Υπάρχει συνένεση για την έκθεση που μας δίνει την ευκαιρία να σημειώσουμε πρόοδο στην πολιτική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Και ε, εννοείται ότι είναι σημαντική αυτή η συμφωνία. Την ασθενίζομαι λοιπόν και τη στηρίζω. Εγώ με τον συνάδελφο Χόρνας ε, Φερνάντε, κατέθεσα την τροπολογία υπαριθμών 51 που αφορά τα παθητικά υποκείμενα ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι η οδηγία που εγκρίνουμε προβλέπει μόνο η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ε, φορολογικών διοικήσεων να αφορά τους κατόχους ε, των λογαριασμών στις φορολογικές διοικήσεις. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρημάτων που υπάρχει ήδη και λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι τα υποκείμενα αυτής της φορολογικής έρευνας ε, δεν περιορίζεται μόνο στους κατόχους των ε, λογαριασμών. Χθε η κυρία Γιώροβα, η Επίτροπος, ήρθε στην Επιτροπή των Αγράφων του Παναμά και έδωσε απαντήσεις ε, στους ευρωβουλευτές που απαιτούσαν μεγαλύτερη φιλοδοξία και πιο απαιτητική οδηγία για την καταπολέμηση της νομοποίησης όδων από παράνομες δραστηριότητες. Θα πρέπει λοιπόν να μην περιοριζόμαστε μόνο στους ε, ε, δικαιούχου των λογαριασμών, αλλά και στα, επεκτηνόμαστε στου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμβολογράφου, δικηγόρου και να καλύψουμε με γραφεία, διαχειριστές κεφαλαίων, ε, διάφορα καταπιστευματικά, διαχειριστές καταπιστευμάτων. Οι δικαιούχοι λοιπόν είναι πάρα πολλοί και δυστυχώς η οδηγία δεν τους καλύπτει ε, όσα έχει. Βέβαια αυτή είναι η γνώμη μας γιατί πρόκειται για γνωμοδότηση ουσιαστικά. Το Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει την οδηγία εν αναμονή της δικής μας γνωμοδότησης. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να καταθέσουμε και τις δικές μας προτάσεις. Δεν θα ήταν λοιπόν κακό, μάλιστα θα ήταν σκόπιμο στη γνωμοδότηση του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει, να πετήσει η ανταλλαγή πληροφοριών να μην περιορίζεται μόνο στους ε, κατόχους, ίσως ε, αναφέρονται ως δικαιούχοι των λογαριασμών, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους ε, φορείς των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο τον λόγο. Ναι, κύριε Τσάνη, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Δύο λεπτάκια μόνο και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Για αυτή την εκθέση θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Θεωρούμε ότι η δουλειά του ήταν πάρα πολύ καλή τόσο όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες αλλά και όσον αφορά το κείμενο. Πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός, προς τη διαφάνεια και προς την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οπότε σίγουρα είναι ένα θετικό στοιχείο και ελπίζουμε ότι η αυριανή ψηφοφορία θα έχει θετικό αποτέλεσμα, διότι πραγματικά το περιεχόμενο είναι ύψης της σημασίας και θεωρούμε ότι επιφέρουν βελτιώσεις και ε, κατά τη δική μας άποψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αν δεν ζητάει κανείς άλλο τον λόγο, κύριε Σιγητά, θα θέλατε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος, διότι ουσιαστικά διαπιστώνουμε με χαρά αυτή την ομοφωνία μεταξύ μας. Είδατε τι είπε ο κύριος Τζάινι αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι ένα μικρό βήμα. Ναι, αληθεύει. Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτή τη στιγμή ε, ε, δημιουργούμε επανάσταση ε, στη φορολογία στην Ευρώπη με μια έκθεση, αλλά με μικρά μικρά βήματα θα καταλήξουμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα. Αυτό το μεγάλο βήμα που αναμένουν από εμά οι ε, Ευρωπαίοι ψηφοφόροι. Τα επιχειρήματα που ανέφερε ο κύριος Αγγή για μένα είναι πολύ σημαντικά, έθεσε σημαντικά ζητήματα και ελπίζω ότι αύριο θα επιτύχουμε ε, την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία, ώστε να δείξουμε και στα άλλα θεσμικά όργανα ότι το Ευρωκοινοβούλιο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ε, στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για αύριο. Ναι, αύριο. Και περνάμε στο επόμενο θέμα. Δεν βλέπω όμως την εισηγητριά. Ε, τι ώρα το είχαμε πει. Σε πέντε λεπτά. Μάλιστα. Πέντε λεπτά διάλειμμα λοιπόν. Δεν περιμένουμε την εισηγήτρια. Ε, εντάξει, εννιάμιση το είχαμε πει, έχει τα δίκαια της. Five minutes suspension. So we start. Λοιπόν, ξεκινάμε με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, το οποίο είναι Τραπεζική Ένωση, έκθεση 2016. Ντανούτα Χίμπνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στην έκθεση αυτή αποφάσισα να ομαδοποιήσω τα ζητήματα ανάλογα με τον πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης που αφορούν Νομίζω πως έτσι είναι λογική η δομή. Γι' αυτό ακριβώς ε, έχω βάλει την διάσωση, την λύση και την ασφάλεια καταθέσεων και έχω ξεχωριστό ζήτημα το θέμα του δημοσιονομικού φρένου, το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να είναι ξεχωριστό ζήτημα λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του. Και δεύτερον, επειδή το ζήτημα αυτό ανήκει σε ένα διαφορετικό νομικό πλαίσιο και πρέπει να το δούμε χωριστά. Ίσως θα θυμάστε ότι στα εκτιμώντας ε, της ε, διακυβερνητική συμφωνίας για το ενιαίο ταμείο διάσωσης είχαμε αναφέρει κάποιο δημοσιονομικό αποθεματικό και υπάρχει ήδη, υπάρχουν ήδη κάποιες πιστοτικές γραμμές μεταξύ των κρατών μελών και του ταμείου αυτού. Αλλά ο μηχανισμός αυτός στήριξης ε, θα είναι μεταξύ του ESM και των ε, κρατών μελών. Οπότε θα περάσει και μέσω μιας διακυβερνητικής συμφωνίας μάλλον. με αυτό μάλλον πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση γιατί τα επόμενα χρόνια μάλλον δεν θα περάσει μέσα από την τακτική νομοθετική διαδικασία για την υποπτία τώρα. Θεωρώ ότι το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει γιατί χρειαζόμαστε κατεπηγόντως κάποια δράση εκεί και για να βελτιωθεί το πλαίσιο της ε, χρεοκοπίας, ε, της αφαιρεγγιότητας ε, στα κράτη-μέλη, αλλά και για να τονώσουμε την ανάπτυξη, για να έχουμε λιγότερα δάνεια τα οποία δεν θα εξυπηρετούνται. Μετά το άλλο θέμα, το οποίο είναι σημαντικό, σε σχέση με την εποπτεία είναι ζητήματα που αφορούν την οριστικοποίηση της Βασιλείας Τρία ή όπως και αν το πούμε εν περιπτώσει και ειδικά το πόσο δεσμευτικές θα πρέπει να είναι οι διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. Γι' αυτό αναφέρω αυτά τα ζητήματα στην πρότασή μου. Και προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να στοχεύσουμε στο πλαίσιο αυτό να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού και αυτό το οποίο συμβαίνει στο διεθνές επίπεδο πρέπει να το ακολουθήσουμε, ότι πρέπει να σεβαστούμε δηλαδή αυτή την αρχή, αλλά θα υπάρχουν και κάποιες καταστάσεις όπου ίσως φοβόμαστε ότι οι διεθνείς κανόνες δεν ταιριάζουν στις ανάγκες μας, οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους επηρεάσουμε εν τη γενέση τους όταν γράφονται, όταν καταρτίζονται στο διεθνές επίπεδο, αντί να αποκλίνουμε στη φάση της ε, μεταφοράς ε, στο δικό μας δίκαιο. Για τα εσωτερικά μοντέλα τώρα εστιάζω ιδιαίτερα στην ανάγκη να γίνουν συγκρίσιμα Αλλιώς θα γίνει η ζωή των υποπτικών αρχών πάρα πολύ δύσκολη, οπότε ακριβώ τα οι υποπτικές αρχές έχουν μεγάλη σημασία. Εδώ πέρα αυτό το ζήτημα θίγω. Δηλαδή πρέπει να μην υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλομορφία, να υπάρχει μια τυποποιημένη προσέγγιση και ένα αξιόπιστο πλαίσιο αυτό έχει μεγάλη σημασία, αλλά αναφέρω και το θέμα του ύψους ε, του ισολογισμού ως μια πολύ σημαντική πληροφορία στο πλαίσιο αυτό και κάτι το οποίο νομίζω πως πρέπει να ξαναπούμε εδώ είναι στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Βασιλείας είναι να μην αυξάνονται οι κεφαλαϊκές απαιτήσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να μείνει στην έκθεση και το τρίτο στοιχείο υπό ε, τον πυλώνα της εποπτείας είναι να επανέλθουμε στις ε, συστάσεις της προηγούμενης έκθεσης σε ζητήματα που ακόμα δεν έχουν έλθει στην μεταρρύθμιση του κανονισμού για την κεφαλαιακή επάρκεια, τις κεφαλαιακές απαιτήσει και βεβαίως ε, τα ζητήματα τα οποία είχαμε πέρσι για τις εθνικές επιλογές και τη διακριτική ευχέρεια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κάνει πάρα πολλά εδώ, αλλά νομίζω πως τώρα επαφίεται στην Κομισιόν να αναλάβει και να δει ε, τι μπορεί να γίνει αυτόματο και τι πρέπει να διαγραφεί. Οπότε τονίζω την ανάγκη να υπάρξει κάποια εναρμόνιση για να διατηρηθεί η ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς. Θα ήθελα λοιπόν οι συστάσεις αυτές να επαναληφθούν. Το τρίτο και σημαντικό είναι η προληπτική αυτή αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους και της σχετικής έκθεσης θα πρέπει νομίζω να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση και βεβαίω υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αλλάξει η αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους. Ξέρουμε πως η Επιτροπή της Βασιλείας ασχολείται εδώ και καιρό με αυτά. Οπότε ίσως το έξυπνο θα ήταν να περιμένουμε να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα πάνε αυτές οι συστάσεις, αλλά θα πρέπει να έχουμε και δική μας άποψη. Τώρα για την ε, λύση των τραπεζών, την εξηγένση, νομίζω πως μόνο το Βέλγιο ακόμα δεν έχει δημοσίευσει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δικαίωμα δεν ξέρω, αλλά κατά βάση έχει ολοκληρωθεί και εκεί η διαδικασία και εκεί πέρα αξίζει να αναφέρουμε κάποια ζητήματα. Πρώτα από όλα τα ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή ενός νέου πλαισίου για να υπάρξει αξιοπιστία, αλλά και αυτό το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό σήμερα, η ε, αλληλεπίδραση με το καθεστώς ε, των ε, κρατικών ενισχύσεων γιατί ο στόχος βεβαίως του συστήματος αυτού ήταν ακριβώς ε, να τελειώσει επιτέλους το ότι πάντα πληρώνουν οι φορολογούμενοι όταν χρεοκοπεί μια τράπεζα. Οπότε πρέπει να το δούμε από την πλευρά των κρατικών ενισχύσεων. Μετά. Α, να τελειώσω, ναι. Στην περίπτωση λοιπόν της εξυγένσης κοιτάω ακριβώς ποια είναι η ιεραρχία των πιστωτών, να υπάρξει μια εναρμόνιση και πρέπει να δούμε και τους ε, τρόπους ακριβώς κατάταξης ε, και προτεραιότητας του χρέους, ειδικά εφόσον είπαμε ότι η συμβατική τέτοια δεν είναι η καλύτερη και θα πρέπει να πιέσουμε το Συμβούλιο να καταλήξει σε μια κοινή προσέγγιση. Και το τελευταίο θέμα για την εξυγένση είναι το θέμα της μεταφοράς των προδιαγραφών της ΤΙΛΑΚ και των σχετικών ζητημάτων για να μπορέσουμε να συμβάσουμε τις, ε, την BRD, την TILAC, ε, τη συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών δηλαδή. Θα πρέπει λοιπόν να μην ε, προδικάσουμε τίποτα, να μην προκαταλάβουμε την νομοθετική έκθεση, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι θα έλεγα γενικές ανησυχίες και συμφωνήσαμε κατά διάρκεια της πρώτης ε, συνεδρίασης με τους κοιοδησίγητες ότι θα πρέπει να μπει στην έκθεση ένας πίνακας που θα συγκρίνει τις ε, συστάσεις που έγιναν πέρσι και τις ε, δράσεις της Κομισιόν να υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια να εξετάζουμε το πώς υιοθετούνται οι συστάσεις μας ή δεν υιοθετούνται αναλόγως αλλά επίσης θα υπάρχει έτσι και πραγματική αξία στην δουλειά μας. Και εδώ τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και με συγχωρείτε αν μακρηγόρησα. Thank you. Σας ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα τους σκιώδεις ηγητές. Κυρία Ντελβό, σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω πρώτα την Τάνωτα Χίμπνερ, την εισηγητριά μας, και να τη συγχαρώ μαζί με τους ε, βοηθούς του επιτελείου και τη γραμματεία για την ε, πολύ αξιόλογη έκθεση που έχει πολύ σαφή δομή, είναι ευανάγνωστη και άπτεται πολύ σημαντικών ε, ζητημάτων της Τραπεζικής Ένωσης. Μάλιστα συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα είπε η συγγήτρια και συμμερίζομαι τις εντυπώσεις που αποκόμισε σε σχέση με την πορεία αυτή της θέσπισης της Τραπεζικής Ένωσης, χωρίς όμως να υποβαθμίζω ή να υποτιμώ την πρόοδο που έγινε, θα ήθελα να δηλώσω ότι κατά τη γνώμη μου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η Τραπεζική Ένωση. Θα πρέπει να σημειώσουμε και άλλη επιπλέον πρόοδο, για παράδειγμα στο σημείο Α λέει ότι έχει θεσπιστεί η Τραπεζική Ένωση, αλλά δεν συμφωνώ πλήρω με αυτή τη διαπίστωση. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι πλήρης ακόμη η Τραπεζική Ένωση. Τώρα, έχω και με άλλες δύο επιστώσεις σας διαφωνώ. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε κάποια μέτρα για τη μείωση του κινδύνου, αλλά δεν συμφωνούμε με την καθυστέρηση ε, στη θέσπιση ε, αυτή. Γιατί μια σταθερή τραπεζική ένωση χρειάζεται και έναν τρίτο πυλώνα. Και αν έχουμε καθυστερήσεις ε, στα ίδια ουσιαστικά καθυστερούμε τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και κάποια άλλα θέματα ίσονος σημασίας ε, και θα καταθέσω και τροπολογίες για τη διάδραση μεταξύ, την αλληλεπίδραση μεταξύ ευρωπαϊκών αρχών και εθνικών αρχών. Επίσης, θέλουμε να ενισχύσουμε τη μακροπροληπτική εποπτεία και επίσης υπάρχει το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που γίνεται όλο και πιο επίγον και σημαντικό. Είχαμε μια συνεδρία στους σχεδόν εισηγητών και συμφωνώ με τις προτάσεις του Σβέν Κίγκολτ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε δελεχώς και την περσινή έκθεση ώστε να έχουμε μια συνέχεια στην επισκόπηση και τον απολογισμό των εξελίξεων στην Τραπεζική Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν η δική μας έκθεση να είναι η συνέχεια της περσινή ετήσια έκθεση και γι' αυτό χρειάζεται ενδελεχή ανάλυση της προηγούμενης έκθεσης. Επίσης, για το χρονοδιάγραμμα. Έχει παραταθεί κατά μία μέρα η διορία για την υποβολή τροπολογιών αναμένοντας την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρότυπο ΤΙΛΑΚ, τη συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε την έκθεση πριν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να μην μείνουμε πίσω. Γι' αυτό διαρωτώ με πώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα για τις συζητήσεις και την υποβολή τροπολογιών. Αυτά και προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με την εισηγητρία και τους και εισηγητές. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπεντ Λούκε για το ECR. Ο κύριος Λούνς ε, είναι ο δικός μας και οδησηγητής. Ε, λυπάται που απουσιάζει. Θα διαβάσω τη δική του δήλωση. Ο κύριος Λούνας ε, ευχαριστεί την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης και θεωρεί ότι, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες, ότι κάποια στοιχεία τουλάχιστον είναι θετικά. Ε, το ECR θέλει αλλαγή στην δομή όμως της έκθεσης, γιατί η δομή στηρίζεται στις, στους τρεις πυλώνες της τραπεζικής έκθεσης και είναι λογικό. Βέβαια, η διαφορά σχέση με την περσίνη έκθεση είναι το ξεχωριστό τελευταίο τμήμα που έχουμε για τη δυνατότητα μιας, ενός κοινού δημοσιονομικού μηχανισμού διασφάλισης. Το θέμα του backstop ε, στηρίζεται με το δεύτερο, ε, σχετίζεται με το δεύτερο πυλόν, άρα θα πρέπει να μείνουμε στους, στα τρία τμήματα, τους τρεις πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης και το δημοσιονομικό μηχανισμό προστασίας να το βάλουμε όπως και στην περσινή έκθεση στον ενιαίο αποπτικό μηχανισμό. Επίσης, οποιαδήποτε μορφή δημοσιονομικού μηχανισμού ασφαλείας αγνοείται το γεγονό ότι ε, τα βασικά δημοσιονομικά και φορολογικά μέτρα με βάση τις συνθήκες ε, και χάρη στην επικουρικότητα λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Οπότε, αν τα κρατημέλη θέλουν να, ε, να θεσπίσουν δικό τους μηχανισμό, δημοσιονομικό μηχανισμό διασφάλιση, θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν. Σε ό,τι αφορά το πρώτο πυλώνα, κρίνουμε ότι δεν αφιερώνεται ιδιαίτερη παράγραφος ε, στα, στις προσωμιώσεις ακραίων ε, καταστάσεων, όπως επισήμανε η έκθεση αρχές του χρόνου. Γι' αυτό θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες. Επίσης, ε, συμφωνεί με τη διατύπωση για την έκθεση σε δημόσια χρέος. Θα πρέπει να ενισχυθεί. Επίσης, το θέμα των εξυπηρετούμενων δανείων και του too big to fail. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο πυλώνα, αναγνωρίζουμε την ισορροπημένη διατύπωση τη συγκεκριτρίας. Θα προτιμούσαμε όμω ε, πολύ πιο ισχυρή και αυστηρή διατύπωση και θα επανέλθω στο θέμα αυτό στη συζήτηση που θα γίνει αργότερα για τα έντας. Ο Ισκιώδης ηγητής προσβλέπει σε επικοδομητική συνεργασία φυσικά με την εισηγήτρια και τους σκιώδης ηγητές για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Για την ομάδα ALDE. δεν βλέπω να βρίσκεται εδώ ο μιλητή. Περνάμε στην ΚΟΕ. Ο κύριος Παπαδημούλης, παρακαλώ. you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο σκιώδης ηγετής μας ο κ. Μακαρθή δεν είναι εδώ και έτσι μου ζήτησε να παρουσιάσω εγώ τη δική μας προσέγγιση. Ευχαριστούμε ε, την η δομή της έκθεσης παρέχει τη δυνατότητα να επιταθούμε στα διάφορα στοιχεία της Τραπεζικής Ένωσης και στην εξυγίανση. συμφωνούμε με το ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα too big to fail κατά την άποψή μας είναι ένα σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να έχει κυρίαρχη θέση στην έκθεση. Δεν αποτελεί απλά θέμα εποπτείας, είναι συστημικό πρόβλημα ενώ η συγκεκριά αναφέρεται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με μη συγκεκριμένο τρόπο, ελπίζω ότι στην τελική εκθεσή θα υπάρχει μια πιο λεπτομερή ανάλυση των αιτιών του προβλήματο αυτού και θα υπάρχουν και κάποιε προτάσει λύσεων. Κατά την άποψή μα, ε, ω την ετήσια εκθέση θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια ανάλυση των βασικών εξελίξεων στον πραγματικό κόσμο του τελευταίου έτου που επηρεάζουν την υλοποίηση τη Τραπεζική Ένωση. Θα πρέπει επίση να συμπεριλαμβάνεται ο τρόπο με τον οποίο εγκαθιδρύεται ο μηχανισμό που θα οριστεί στο πλαίσιο τη Τραπεζική Ένωση για προσαρμογή σε αυτέ τι εξελίξει στον πραγματικό κόσμο. Α πάρουμε το παράδειγμα τη Deutsche Bank. Άριστο παράδειγμα αποτυχία αντιμετώπιση του ζητήματο του Big to Fail και της ε, μεροληπτικής αντιμετώπισης των διαδικασιών της ε, ΕΚΤΑ. Η Deutsche Bank είναι ο βασικός παράγων συστημικών κινδύνων παγκοσμίω. Και οι Financial Times περιγράψαν την τράπεζα αυτήν ως δομικά αδύναμη με 1,8 τρισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τις εμπορικές της δραστηριότητας, γεγονός που δείχνει τους κινδύνους μη αντιμετώπιση του προβλήματος του Big to Fail των μεγάλων συστημικών τραπεζών και των τεράστιων εκθέσεων σε παράγωγα. Εμείς προτείνουμε τη διάσπαση των μεγάλων τραπεζών και τη διαχωρισμό των επενδύσεων και των εμπορικών δραστηριοτήτων των τραπεζών ως μοναδικό αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος με το ενδεχόμενο μιας ε, επερχόμενης ε, τραπεζικής κρίσης ξανά θα ε, γίνει μια ακραία δοκιμή, θα δοκιμαστούν οι συστημικές τράπεζες. και δεν ξέρουμε αν με τα μέσα που έχουμε αυτή τη στιγμή θα καταφέρουμε να αποτρέψουμε την κατάρρευση μιας μεγάλης Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Η Τραπεζική Ένωση επίσης παρέχει περισσότερες εξουσίες σε μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν έχει μεταρρυθμιστεί. Συνολικά όπως έχει η Τραπεζική Ένωση σήμερα είναι απίθανο να μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια ε, εκτεταμένη ε, τραπεζική κρίση αποτελεσματικά και το Κοινοβούλιο πρέπει να το αναγνωρίσει αυτό. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την εκθέση αυτή ώστε να επισημάνουμε τις απόψεις των βουλευτών και να διαμορφωθεί μια απόκριση ε, σε, στις διάφορες εξελίξεις ε, στον τραπεζικό τομέα. Ευχαριστούμε, Σπαγγίγκλη, για τους πρασίνους. Είναι λίγο περίεργη αυτή η συζήτηση. Αλλά καμιά φορά πρέπει να συμβαίνουν και περίεργα πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η δομή και τα ζητήματα που αναλύει ο εισηγητής είναι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε και τώρα έχουμε μια καλή βάση για να το γεμίσουμε με λίγο επιπλέον περιεχόμενο και πολλά από τα πράγματα που είπαμε στην περσινή έκθεση εξακολουθούν να ισχύουν και κατά την άποψή μου και για τις συζητήσεις που είχαμε σήμερα πρέπει να δούμε ξεκάθαρα πως ένα χρόνο μετά την τελευταία μας έκθεση έχουμε απαντήσει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και όταν βλέπουμε την έκθεση της ε, Κομισιόν, στην περσινή δική μας έκθεση, βλέπουμε ότι διαλέγουν ό,τι τους βολεύει. Δηλαδή απαντάνε στα ζητήματα που θέλουν και απλά γνωρούν αυτά που δεν τους αρέσουν. Και ή θεωρούν ότι δεν είναι σε θέση να απαντήσουν. Πρέπει όμως να παίρνουμε τον εαυτό μας στα σοβαρά. Οπότε βασικά πρέπει να επανέλθουμε σε όλα τα εισδήματα τα οποία δεν είδαμε σωστά και ελπίζω η γραμματεία να το κάνει αυτό για αυτή την έκθεση αλλά και για άλλες εκθέσεις. Ε, έχουμε την έκθεση Γκουλάρ, ε, πάρα πολύ παρόμοια ε, για την Βασιλεία και για άλλα παγκόσμια θεσμικά όργανα. Επίσης για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και εκεί πέρα απαντούσαν σε ό,τι ήθελαν. Πρέπει να έχουμε μια πιο συστηματική προσέγγιση και να φροντίσουμε να απαντάει η Κομισιόν και να δούμε μετά που βρισκόμαστε και να μην ξεκινάμε από το μηδέν σαν να μην ε, είχαμε ξανακάνει τίποτα στο παρελθόν. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω την γραμματεία και θα ήθελα να παρακαλέσω τους αδέλφους να είμαστε πιο συστηματικοί. Επί της ουσίας, Έχουμε κάποια νέα ζητήματα σε σχέση με την περσινή έκθεση, παραδείγματο χάρη για τα τεστ κοπόσεως αυτά είδαμε πως υπήρξε ειδική μεταχείριση της Deutsche Bank. Αυτό δεν πρέπει να το δεχτούμε. Υπήρχε και εθνική διακριτική ευχέρεια για άλλες τράπεζες. Έχω την εντύπωση πως η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή έχει περιορισμένες αρμοδιότητες για να ελέγξει την εθνική διακριτική ευχέρεια στα στρες τεστ αυτά και θεωρώ ότι πρέπει να ότι έχουμε πραγματικά συμφέρον να είναι ενιαία αυτά τα stress test. Δεύτερον, έχουμε ένα πρόβλημα διαφάνειας που δεν είναι παντού ίδια. τράπεζες αυτές ε, που ήταν αρμοδιότητα της CBA πραγματικά είχαν μεγάλη διαφάνεια, αλλά οι τράπεζες όπου ήταν εσωτερικής διαδικασίας της ΕΚΤ δεν είχαν καθόλου διαφάνεια, οπότε υπάρχει μια άνηση μεταχείριση και νομίζω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν με έναν τρόπο ευρωπαϊκό με τον ίδιο τρόπο για όλους και για όταν μιλάμε για την διακριτική ευχέρεια και την διαφάνεια. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο νομίζω πρέπει να θίξουμε πολύ περισσότερο, είναι ε, το οικονομικό έγκλημα και η έλλειψη προστασίας των καταναλωτών. Ξέρουμε ότι έχει περιορισμένη εντολή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι φυσιολογικό οι τράπεζες ε, που έχουν σοβαρά προβλήματα με το οικονομικό έγκλημα να μην το πληροφορείται καν η υποπτική αρχή. Και το ίδιο έχουμε δει με την προστασία των καταναλωτών. Έχουμε λοιπόν αυτό το πλαίσιο της εξυγίανσης των τραπεζών, αλλά αντιμετωπίζουμε πολιτικά προβλήματα όταν ε, κάποια στοιχεία ενεργητικού είναι στα χέρια ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, όπως έχουμε δει με τις Ιταλικές τράπεζες. Και άρα υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση του πλαισίου εξυγένσης με την προστασία των καταναλωτών. Πέρσι η κυρία Κιόνικ μας υποσχέθηκε έναν κατάλογο των προβλημάτων στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν έχει ακόμα εκπληρώσει την υπόσχεσή της. Και θέλουμε το σύστημά μας ε, εξυγένσης των τραπεζών να είναι αποτελεσματικό και εξακολουθώ να πω πως υπάρχουν προβλήματα για την συμμετοχή στην διάσωση κάποιων στοιχείων του ενεργητικού και υπάρχουν τάσεις να πάει η παραγωγή των, δημοσιο... των χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες γιατί ελπίζουν ότι εκεί θα είναι δυσκολότερο το Μπέιλιν. Ε, ελπίζω αυτό να μην είναι αποδεκτό και τελικά θα μπορέσει να δώσει περαιτέρω πλεονεκτήματα στους φορολογικούς παραδείσους. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε καλή συνεργασία με ολόκληρο την κοινοβούλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάρκο Βαλή. Ναι, ευχαριστώ. Θα μιλήσω εκ μέρους του σκιώδου του Μάρκο που δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Συγγήτρια πολλές ευχές για μια καλή συνεργασία κατά τις συζητήσεις και για τις τροπολογίες. Πιστεύω όμως ότι απομένει πολλή δουλειά να γίνει κατά την απόψή μας για αυτή την έκθεση. Ξεκινώντας από ένα σημείο, όταν διαβάζω αυτό που υπάρχει εδώ στην έκθεση ε, και κοιτάζοντας ταυτόχρονα τη σημερινή κατάσταση του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη, βλέπω ένα χάσμα μεταξύ της θεωρίας, ε, της γραπτής θεωρίας και της πραγματικότητας των γεγονότων και κατά την απόψη μου αυτή η έκθεση θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία να πούμε καθαρά τι δεν λειτουργεί σωστά στο, ε, πρόγραμμα, στο σχέδιο της Τραπεζικής Ένωσης, τι δεν λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια, διότι σίγουρα κάποια πράγματα δεν λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε ή λειτουργήσαν άσχημα και οι επιδόσεις του τραπεζικού συστήματος, οι δυσκολίες που δεν αφορούν μόνο ορισμένους τομείς ή ε, ε, ορισμένες περιοχές ε, αλλά έχουν διαδοθεί αρκετά, είναι πλέον ορατές σε όλους. Είναι κρίμα που δεν υπήρξε κάποια κριτική όπως αυτή του μηχανισμού εποπτείας, του νέου μηχανισμού εποπτείας που ε, τους τελευταίους μήνες εργασίας του έχει αναδείξει πολλά κενά ότι δεν μπορεί να καθορίσει και να εντοπίσει με τρόπο επαρκή τους κινδύνους που ενέχει αυτή τη στιγμή στους προπολογισμού του το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Δεν ακούγεται κάποια επικοδομητική κριτική ε, όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των stress test και της αναθεώρησης ποιότητας. Απομένουν και δύο θέματα πρέπει να αναλυθούν λεπτομερώς ε, θέματα όπου ανέδειξαν αποτυχίες ε, τα stress test, οι κίνδυνοι της αγοράς που κατά την άποψή μου δεν λαμβάνονται παρκώς υπόψη από την ανάλυση του SSM και της EBA και οι νομικοί κίνδυνοι που όπως είδαμε στην περίπτωση της Deutsche Bank θα μπορούσαν να, ε, να λάβουν τεράστιες διαστάσεις και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος θέτοντα σε κίνδυνο ολόκληρο το σύστημα ουσιαστικά διότι μιλάμε για πολύ σημαντικά ποσά. Δεν ακούγεται ισχυρή κριτική για το μοντέλο της BRRD που κατά την απόψή μου έδρασε αντίθετα από ό,τι έπρεπε. Δεν εξαλείφθη τους κινδύνους bailout που παραμένουν ε, ισχυροί, δεν εξαλείφει τους κινδύνους ε, συμμετοχής ε, των συμμετεχόντων για τις διασώσεις των τραπεζών και κυρίως δεν καθιστά το τραπεζικό σύστημα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα πιο σταθερό. Αντιθέτως, το καθιστά πιο αβέβαιο, λιγότερο σταθερό. Αυτό είναι ένα σημείο ε, το οποίο θα πρέπει να αναλύσουμε σε περισσότερο βάθος κατά την απόψή μου και από την απόψη της αποτελεσματικότητας της οικοδόμησης αυτού του buffer των ε, αξιών ε, που χρησιμοποιούνται για τον Μπέιλιν. Και κάτι τελευταίο που ανέφεραν και κάποιοι συναδελφοί, το γεγονό ότι η Τραπεζική Ένωση σήμερα έτσι όπω έχει δημιουργηθεί δεν επιλύει το πρόβλημα του too big to fail των τραπεζών που είναι πολύ μεγάλε για να αποτύχουν. Ε, από αυτή την άποψη θα πρέπει να απαιτηθεί ισχυρότερη δράση, ε, κυρίως στο ζήτημα της μόχλευσης εντός του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, που παρότι έχει μειωθεί μετά από την κρίση του 2008-2009 για ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα παραλαμμένει ένα ισχυρό παράγον και πιστεύω ότι θα πρέπει να δράσουμε και σε αυτό το θέμα. Τώρα όσον αφορά το τελευταίο σημείο, το σύστημα ε, κοινών εγγύσεων και ασφαλίσεων για των καταθέσεων που θα έπρεπε να αποτελεί το πυλώνα που θα συμπληρώσει, θα ολοκληρώσει την Τραπεζική Ένωση και για το οποίο θα συζητήσουμε αργότερα μέσα στη σημερινή μέρα. Πιστεύω ότι για αυτό το θέμα χρειάζεται κάποιος προβληματισμός να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος κατά την οικοδόμηση της Τραπεζικής Ένωσης και να φτιάξουμε ουσιαστικά ένα εργαλείο το οποίο θα μειώνει τους κινδύνους του τραπεζικού συστήματος που θα καθιστά το τραπεζικό ε, σύστημα πιο σταθερό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος και μεγάλος κατά την άποψή μου να δημιουργήσουμε ένα ε, μόρφωμα ε, το οποίο θα επιτύχει τον αντίθετο στόχο, δηλαδή ουσιαστικά θα γεννήσει ένα ποντικάκι το οποίο θα αποσταθεροποιήσει ολόκληρο το σύστημα. Αυτά θα είναι τα ζητήματα στα οποία θα επικεντρωθούμε εμεί στις δικές μας τροπολογίες. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω τον ομιλητή του ΙΕΝΕΦ, οπότε ξεκινάμε το Catch και δίνω το λόγο στον εαυτό μου για την τρίτη παρέμβαση. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, την κυρία Ντάνοτα Χιούμπνερ, για την έκθεσή της Πιστεύω ότι η έκθεση είναι αξιόλογη και συμφωνώ με πολλά σχόλια. Απ' την άλλη πλευρά και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό δημοκρατικό σώμα που κάνει τον απολογισμό αυτού του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε πολύ πιο κλεπτισμένο ελεγκτικό έργο. Και συμφωνώ ότι υπάρχουν πολλά επιμέρους ζητήματα που μπορεί να μην είναι πρωταρχική σημασία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τα παραμελήσουμε. Δηλαδή, το θέμα των ε, λειτουργικών επιχειρησιακών ζητημάτων, ε, διοικητική κατανομή αρμοδιοτήτων, τρόπος με τον οποίο JSD ε, ασχολείται με τις τράπεζες, το χρονοδιάγραμμα, αποφυγή διπλών εκθέσεων. και κατά πόσο θα λαμβάνεται υπόψη η αναλογικότητα στον έλεγχο. Έχουμε άλλα θέματα επιμέρους ε, πολύ επίσης ε, σημαντικά που αποφασίσαμε να ενταχθούν στον Δημοκρατικό Κοινοβουλευτικό Έλεγχο. Δεν θα λέω ότι θα πρέπει να δώσουμε συνέχεια στο παραμικρό ζήτημα, αλλά καλό θα ήταν να έχουμε μια πολύ έκθεση και να δώσουμε συνέχεια σε πολλά από αυτά τα επιμέρους θέματα. Τώρα για ένα πολιτικό θέμα. Πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερη ευάθυνση στο θέμα της ε, ε, ικανότητας ε, του επαρκούς επίπεδου εποπτικής στρατηγικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κατάλληλο επίπεδο ολοκλήρωσης των γενικών διευθύνσεων που ασχολούνται με επιμέρους στοιχεία των τραπεζών και μια οριζόντιας ολοκλήρωσης. Αυτό το επισημάναμε και στην προηγούμενη της έκθεση. Για παράδειγμα, τι θα πει η εποπτική στρατηγική πρόβλημα κερδοφορία. Ε, χρειάζεται μεγαλύτερη εξυγίαση του κλάδου. Μερικέ φορέ όμω έχουμε την εντύπωση ότι υιοθετούμε διαφορετικέ προσεγγίσεις οι διάφορε, επιμέρου ε, γενικέ διευθύνσει. Άλλοι επικεντρώνονται στην εξυγίαση, άλλοι στην ε, πρόληψη, άλλοι στην επάρκεια κεφαλαίων και ίσως δημιουργηθεί δοθεί εντύπωση ότι είναι αντικρώμενες αυτές οι προσεγγίσεις. Χρειάζεται λοιπόν μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση και συνάφεια. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Και όλα τα θέματα τη αναλογικότητα επίση που επισημάναμε. Σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα, έγινε μεταρρύθμιση, έγινε μια διευκρίνηση. Είτε μα αρέσει είτε όχι. Εγώ θεωρώ ότι είναι σκόπιμη και θα πρέπει να το τονίσουμε γιατί ήταν ένα από τα σημεία που είχαμε ζητήσει εμείς, κατευθυντήρες γραμμές για το δεύτερο πυλώνα. Και, και για το θέμα του ΜΡΕΛ, για την ελάχιστη απέτηση ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, θα πρέπει να κρατήσουμε την ίδια προσέγγιση. Και επίση το, επίπεδο δημοσιοποίηση κάποιων στοιχείων. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των κατευθυντηρίων γραμμών και των απαιτήσεων. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, επίση συμφωνώ με τον Σβέν Γκίγκολτ και επίσης ε, θέματα μακροπροληπτικής εποπτείας. Ε, καλό θα ήταν ε, να μην παραμείνω εδώ και να δοθεί και κάποια συνέχεια. Σε ό,τι αφορά το πλάνο της εξηγήση. με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού μιλήσαμε για τη ερμηνεία της παρούσας οδηγίας για την εγγύηση καταθέσεων. Είναι σημαντικό λοιπόν να ζητήσουμε αντιμετώπιση του προβλήματος με μία άμεση λύση για να γίνει ε, εύχριστη αυτή η πρόταση του νομοθέτη για να μην χρησιμοποιηθούν κάποια συστήματα εγγύης καταθέσεων ως ε, κρατικές ενισχύσεις. Επίσης έχουμε ένα δεύτερο στρώμα εθελοντικό για να αποφύγουμε και την επικάλυψη που θα ήταν αντιπαραγωγική και ίσως σε αυτή την έκθεση θα μπορούσαμε να βάλουμε και αυτό το θέμα. Ίσως καταθέσω και σχετική τροπολογία. Τέλος, για το, την έκθεση δημόσιο χρέος. Συμφωνώ ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί με τέτοια έκθεση ως ασφαλές περιουσιακό στοιχείο. Και θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και ως προς τα μέτρα που θα πρέπει να παίρνουν κάποιο τεστ κόστους οφελους και την ίδια ε, επιφύλαξη και πρόληψη θα πρέπει να δείξουμε γενικώ. Να έχουμε μια ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους των επιμέρους μέτρων που θα προταθούν. Θα πρέπει πρώτα τα μέτρα να περάσουν το τεστ κόστους οφελους και μετά να μειώνεται ο κίνδυνος της έκθεσης ε, σε δημόσιο χρέος. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Άλλωστε είναι θέματα που εξετάζονται και στη Βασιλεία. Ίσως θα πρέπει να περιμένουμε την έκβαση των συζητήσεων για το πλαίσιο της Βασιλείας για να οριστικοποιήσουμε και αυτό το σημείο. Πάντως το πνεύμα του κειμένου είναι σωστό, δηλαδή δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα, αλλά ρεαλιστικό. Επόμενος ομιλητής παρακαλώ. No other ε, για το catch the eye. Ωραία, λοιπόν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να, σας, ε, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, που διάβασαν την πρόταση. Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν συντάξει κανείς μια πρώτη εκδοχή έκθεσης έχει κάποιου περιορισμού και πρέπει να αποφασίσει αν θα κινηθεί προ επισήμανση ζητημάτων και όχι εμβάθυνση του, ε, ή αν θα εμβαθύνει σε ένα-δυο ζητήματα χωρί να επεκταθεί ε, και σε άλλα. Εγώ διάλεξα λοιπόν αυτή την προσέγγιση, τη διευρυμένη προσέγγιση πολλών ζητημάτων για να γίνει κάποια συζήτηση. Αλλά εκτιμώ και τα σχόλια φυσικά που ακούστηκαν για την πιθανή επέκταση του αντικειμένου της έκθεσης όπως ε, είπατε, πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτυχουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ του τι ανήκει σε μια έκθεση για Τραπεζική Ένωση που δεν είναι έκθεση της τραπεζικής κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2016, οπότε πολλά είναι τα ζητήματα τα οποία θα χρειαστεί να συζητήσουμε στις ε, συναντήσεις των σχεδόν, δηλαδή πόσο πολύ θα τραβήξουμε την ανάλυση της κατάστασης του τραπεζικού τομέα σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι συμμερίζομαι και συμφωνώ με τα περισσότερα σχόλια όσον αφορά την κατάσταση. Ένα σχόλιο ακούστηκε από το ECR όσον αφορά το σκεπτικό στο οποίο βασίστηκε η προσθήκη αυτού του ζητήματος που ανοίξει το κομμάτι του, της εξυγένσης. Ε, ε, το ζήτημα του κοινού ε, δημοσιονομικού μηχανισμού ασφαλείας πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε και θα πρέπει να αναφερόμαστε πάντα και στους τρεις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την εκθέση. Αλλά κάθε χρόνο μπορεί να προκύπτει ένα άλλο ζήτημα ως εξέχον, ως ιδιαίτερα σημαντικό. Οπότε θα πρέπει να δείξουμε κάποια ευελιξία λοιπόν σε τέτοιες εκθέσεις. Δηλαδή το να συμπεριλάβουμε ένα-δύο ζητήματα τα οποία παρότι ανήκουν στη στενή δομή της ε, Τραπεζικής Ένωσης θα πρέπει να υπογραμμίζονται κάπως με, ε, για να τους κάποιο ξεχωριστό χώρο στην έκθεση. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντική αυτή η συζήτηση. Ένα ζήτημα το οποίο, ε, στο οποίο αναφέρθηκε ο Ρομπέρτο είναι το ζήτημα του να δούμε πώς η διοίκηση της ε, Τραπεζικής Ένωσης και της Εποπτείας ε, λειτουργεί σήμερα. Φυσικά το ανέφερα αυτό, αλλά υπάρχει και η διοικητική οργάνωση του SSM, ε, οι εξουσίες της. Εκεί αναφέρεται το ζήτημα αυτό και πιστεύω ότι το γεγονός του πώς ασκείται η εποπτεία, πώς ασκούνται τα καθήκοντα ε, στο πλαίσιο αυτό της Τραπεζικής Ένωσης είναι κάτι σημαντικό. Έχω αναφέρει τα σχετικά ζητήματα στην έκθεση, αλλά θα μπορούσαμε φυσικά να τα εμβαθύνουμε και περισσότερο. Τώρα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι θέμα του κατά πόσο είναι δυνατό ή όχι ε, να επεκτείνουμε την προθεσμία σε σχέση με την προηγούμενη, να την παρατείνουμε ε, σε σχέση με αυτό που προτάθηκε από την γραμματεία βάσει του φόρτου εργασίας και της όλης διαδικασίας μέχρι την Ολομέλεια που είχε προταθεί αρχικά και μετά είδαμε μήπως μπορούμε να διατηρήσουμε παρόλα αυτά την ημερομηνία ψηφοφορίας για την τελική ψηφοφορία και να παρατείνουμε την, τροπολογία, την προθεσμία ε, τροπολογιών ε, αυτή η παράταση που προτείνεται μας ε, επιτρέπει να μην ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του χρόνου το καλοκαίρι. Καλό είναι η έκθεση αυτή να ψηφιστεί το νωρίτερο δυνατόν στις αρχές του επόμενου έτους και Κάτι επίσης που πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, θα είναι αυτό που θα μας στείλει η Κομισιόν τέλη του μήνα, ελπίζω, για το ΣΕΡΑ και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη καθώς θα μελετάμε τις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Θα λάβουμε υπόψη και αυτές τις επιπλέον πληροφορίες από την Κομισιόν, αλλά μάλλον είμαι κατά της παράτασης της προθεσμίας υποβολής τροπολογιών διότι αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα να ψηφίσουμε σε, εύλογο, σε εύλογη χρονική προθεσμία, αρχές δηλαδή του χρόνου του 2017. Αυτή είναι η απόψη μου. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να έχετε ε, μια καρποφόρο συνεργασία όλοι οι συνάδελφοι μεταξύ όλων των ομάδων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε Τανούτα. Ήμουν με την Κλάουντα και κοιτάζαμε αυτά που λέτε. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε δεν θέλετε να αναβληθούν τα πάντα και ειδικότερα όχι η ψηφοφορία στην Ολομέλεια που έχει προγραμματιστεί αυτή τη στιγμή για το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο. Ωστόσο, εξακολουθώ να πιστεύω ότι διατηρώντας αυτή την προθεσμία θα μπορούσαμε ε, ενδεχομένω να μην έχουμε απαραίτητα στι 8 Δεκεμβρίου την εξέταση των τροπολογιών, αλλά να έχουμε την εξέταση των τροπολογιών αρχέ Ιανουαρίου. Όχι. τέλη Ιανουαρίου είπαμε, λέει η συγκήτρια. Ναι, αυτό είδαμε, λέει ο Πρόεδρος. Κατά πόσο μπορεί να βρεθεί κάποια χρονική στιγμή, θα πρέπει να το τσεκάρουμε φυσικά. Επειδή η προθεσμία Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι, ε, λέει ο Πρόεδρος, για ποιο λόγο ε, θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει μεγαλύτερη παράταση, αλλά φυσικά σέβομαι να πάμε δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι, αλλά καταλαβαίνω και την άποψη του να μην πάμε πιο πέρα από το Μάρτιο όσον αφορά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Οπότε ας κάνουμε ένα τεχνικό έλεγχο. Να πούμε, ας πούμε, ότι έχουμε την ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Μαρτίου Και αν τα καταφέρουμε, τα καταφέρουμε. Και αλλιώ ε, θα, δούμε. Θα προσπαθήσουμε να το πλήσουμε σήμερα όλο αυτό, αν συμφωνείτε. Εντάξει, συμφωνείτε. Ωραία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Παίρναμε στο επόμενο σημείο. Που είναι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 Λοιπόν, μια υπενθύμηση για μια συνεδρία σε αυτή τη βδομάδα που σχετίζεται με την ΕΚΟΝ. Πιστεύω θα τα έχετε λάβει όλα, ε. οπότε δεν χρειάζεται. Ναι. Μπορείτε να διαβάσετε αυτά που λάβατε λοιπόν. Δεν χρειάζεται εμένα να επαναλαμβάνω τι θα κάνουμε αυτή τη βδομάδα τέταρτος πολιτικό ε, τριμερής διαλόγο. για το μήνυμα και φάντα έλαβε χώρα τον Νοέμβριο. Συζητήθηκαν το MMF, τα συστήματα για τους υπαλλήλου, κανόνε οι τύποι του MFF και η σταδιακή εισαγωγή σημειώθηκε πρόοδος και έγιναν κάποιες προκαταρκτικές συμφωνίες για ορισμένα ζητήματα. Ο πέμπτος τριμερής διάλογος θα λάβει χώρα στις 14 Νοεμβρίου. Επίσης είχαμε τον πρώτο τριμερή διάλογο για τον κανονισμό προσπέκτους για τις 27 Οκτωβρίου. Ε, καλύφθηκαν τα νομισματικά κατόφλια, υποχρέωση ε, δημοσίευσης Φιλανδίων για τα εθνικά ε, καθεστώτα. Αυτή η απέτηση λοιπόν για το προσπέκτους, ε, το καθεστώς για τα δευτερόντα ζητήματα, η σύνοψη των προσπέκτους, ε, οι πληροφορίες αποστολής και το γενικό έγγραφο ε, καταγραφής. Ε, σημειώθηκε πρόοδο σε πολλά από αυτά τα ζητήματα και ο επόμενος τριμερής διάλογος προγραμματίζεται για τις 15 Νοεμβρίου. Η σύνοψη των αποφάσεων και των συστάσεων από την συνάντηση των συντονιστών της 12 Οκτωβρίου για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα συμφωνήθηκε ότι οι Κομισιόν και οι εκπρόσωποι των Εθνικών Αρχών θα παρουσιάσουν τις δραστηριότητες του στον τομέα σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής, μελέτη της υλοποίησης της ε, νομοθεσίας επίσης θα απαιτηθεί και πιθανή σύνταξη έκθεσης υλοποίησης θα εξεταστεί ως ενδεχόμενο μετά από τα, από τα προηγούμενα βήματα οι συντονιστές υιοθέτησαν το ημερολόγιο και το χρονοδιάγραμμα για τις συνεδριάσεις των διαφόρων ομάδων εργασίας το 2015 για τις δημόσιες ακροάσεις. Εφόσον εγκριθούν από τη διασκέψη των Προέδρων, οι συντονιστές συμφώνησαν να γίνουν το 2017 ακροάσεις για το CCP, μακροοικονομικές πολιτικές στο πλαίσιο να συνεχού περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων. Αυτό δεν είναι ο τελικός τίτλος, δεν είναι ο οριστικό τίτλο, είναι ο παλιός, θα έχει διορθωθεί την πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων, CCTV, Brexit, Βασίλεια 3 και Βασίλεια 4 για τις αποστολές, ε, το πρώτο εξάμεινο 2017, όχι αυτό είναι όλο το 2017 ουσιαστικά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λονδίνο τον Απρίλιο, αφού ενεργοποιηθεί το άρθρο 50, Βερολίνο, 22 με 24 Μαΐου 9 μέλη, Λισαβόνα 20-21 Οκτωβρίου 9 μέλη ΣΥΜΠΗ και Βασιλεία στο Στρασβούργο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοσίνγκτον και Νέα Υόρκη 16-21 Ιουλίου 7 μέλη Σανγκάι, Πεκίνο, Κίνα 18 με 22 ε, Σεπτεμβρίου 7 μέλη IMF ετήσια συνάντηση Washington 11 με 15 ε, Οκτωβρίου 7 μέλη. Συμφωνήθηκε ότι το επόμενο θέμα θα είναι το PSD 2 για την οικονομική διακυβέρνηση. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή με τα μέλη της, ε, του νεοδιοριστέντο Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Αποφασίσαμε να γίνει το συντομότερο δυνατόν μετά από το διορισμό, αλλά λάβαμε ε, μια επιστολή από το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο που θεώρησαν ότι ήταν πολύ νωρί για να έρθουν εδώ ε, πριν καθορίσουν κάποιε συγκεκριμένε θέσεις. Εγώ λυπάμαι για αυτή την επιστολή διότι η πρόταση να γίνει ένας απολογισμός του χρόνου ε, σε μια συνάντηση δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Εμείς ε, μένουμε στο αίτημά μας να έρθουν εδώ και λυπούμαστε που δεν είναι διαθέσιμα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου να έρθουν εδώ για μια ταλήγη απόψεων στην ΕΚΟΝ. Ε, τώρα, διορισμούς. Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα και την επέκτασή του Πρόεδρος ε, Γενική Αναθεώρηση της Διαδικασίας καμία γνωμοδότηση λόγω χρονικών περιορισμών καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός δημιουργίας θέσεων εργασίας γνωμοδότηση ΓΚΟΕ ελάχιστη οικονομική πολιτική για την αντιμετώπιση της φτώχειας γνωμοδότηση για την Γκουέ επίσης και θα συζητήσουμε ε, τις ε, πρωτοβουλίες ε, τον Νοέμβριο. Συμφωνήθηκε λοιπόν ο εισηγητής να συζητήσει το ζήτημα που ζητήθηκε με την αναφορά και να δούμε ποια θα είναι η ποιότητα τη απαντησή μας για την αναφορά και τώρα σε σχέση με τις παρελθούσε πρακτικές ο κ. Χόιερ, πρόεδρος της ΕΚΤ, θα κληθεί ε, σε ακρόαση στην ΕΚΟΝ. Πάμε τώρα στην έκθεση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας Καταθέσεων. Ο συγγετής μας είναι ο κύριος Λάγκε που κατέθεσε το σχέδιο έκθεσης και θα το παρουσιάσει σήμερα η κυρία Λάγκη, συγγνώμη. εστέριξε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, φαντάζομαι δεν είμαι η μόνη που ε, το μυαλό τη είναι καλυμμένα από άλλα θέματα που δεν αφορούν το ΕΔΙΣ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλεια Καταθέσεων, αλλά τι να κάνουμε. Επίση, 12 ακριβώ πρέπει να φύγω, οπότε καλό θα ήταν να ολοκληρώσουμε μέχρι τότε. Αλλά έχουμε παρόλα αυτά μια μισή ώρα για να συζητήσουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύης Καταθέσεων και Παρόλο που το θέμα είναι επίμαχο, νομίζω ότι μια μισή ώρα αρκεί για τη συζήτηση. Α ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω του και ηγητές ε, για τα σχόλιά του αλλά και για την ε, ευελιξία του και ευχαριστώ και τι υπηρεσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με βοήθησαν πολύ στην εκπόνηση τη έκθεση. Πώ έχει η κατάσταση. Όπω γνωρίζουμε, έχουμε τεχνικό έργο, αλλά πολύ αργή, για να μην πω μηδενική πρόοδο στο Συμβούλιο. Οπότε από εμά εξαρτάται να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το ζήτημα και πολλές ε, πολιτικές ομάδες ε, θεωρούν ότι είναι και το θέμα. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης προσπάθησα να εκπληρώσω διάφορους στόχους. Ο πρώτος και βασικός είναι σε ασφαλιστικές δικλείδες για κάθε καταθέτη στην Ευρώπη, όπου και αν διαμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγγύψει αυτό το θέμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύης Καταθέσεων, όχι από ε, πλευρά τεχνική, αλλά από τη σκοπιά του καταναλωτή, του, του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κοινό στόχο των σκιωδών εισηγητών. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα με λιγότερη έκθεση των τραπεζών. Δεν θα πρέπει ε, καμία χώρα ή κανένα σύστημα αγγής καταθέσεων να, είναι χειρότερο από τα άλλα. Γι' αυτό και θέλουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Περιορισμό του ηθικού κινδύνου επίση, αλλά με τρόπο που να συνδέεται με το σύστημα αγγή καταθέσεων και όχι να χρησιμοποιείται ω πρόσχημα για την έλλειψη πρόοδου. Επίσης, ε, επιμερισμός κινδύνων και μείωση κινδύνων. Αυτό θα πρέπει να είναι αλληλένδετα. Ωραία τα λόγια και εύκολα, αλλά όταν ερχόμαστε στη διατύπωση και στο πώς θα το επιχειρήσουμε, αυτό είναι πιο δύσκολο. Τα έργα είναι πιο δύσκολα από τα λόγια. Και εκεί υπάρχει διάσταση απόψεων, να είμαστε ειλικρινεί. Τελευταίο στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η φιλοδοξία μας να μην έχουμε μία ακόμη ε, διακυβερνητική συμφωνία για το θέμα αυτό. Γνωρίζω ότι δίστανται οι απόψει ειδικά στο Συμβούλιο, για αυτό το ζήτημα, αλλά θεωρώ ότι μία ακόμη διακυβερνητική συμφωνία που δεν εμπλέκει ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Γι' αυτό και υπέβαλα την πρότασή μου ευελπιστώντα ότι θα τύχει υποστήριξη ε, για να αποφύγουμε μια επιπλέον διακυβερνητική συμφωνία. Βέβαια, ε, είναι γνωστό ότι υπάρχει διάσταση απόψεων ακόμη και στην ομάδα μας ε, σε ό,τι αφορά την αρεσιμότητα, το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα της πρόταση αυτής. Για παράδειγμα, ως προς το περιεχόμενο, αν πούμε ότι θέλω αμέσως να περάσουμε στην τελική φάση του ΕΝΤΙΣ, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύηση Καταθέσεων, τότε θα έχουμε περίπτωση τη συζήτηση για την αρισιμότητα, δηλαδή τι προποθέσει θα πρέπει να πληρούνται για να περάσουμε σε αυτή την τελική φάση. Και σε αυτά τα θέματα υπάρχει διάσταση απόψεων. Για μένα το πιο σημαντικό είναι, δεδομένη έλλειψη πρόοδου στο Συμβούλιο, αν μη τι άλλο να δώσουμε το αναρκτήριο λάκτισμα. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε να δώσουμε πνοή σε αυτό το θέμα. Ίσως θα μπορούσαμε να ε, συγκροτήσουμε το έντις γύρω από δύο φάσεις. Καταρχήν ε, να ανα, αναζωογονήσουμε τη φάση της αντασφάλισης που ξεκίνησε το 1999 ε, και ξεκίνησε τουλάχιστον για πέντε χρόνια. Το θέμα της ρευστότητας είναι πολύ σημαντική. Οι περισσότεροι θέλουν άμεση εξόφληση. Βέβαια, ίσως ε, μερικά συστήματα καταθέσεις καταθέσεων δεν θα μπορέσουν να το εξασφαλίσουν. Θέλουμε φιλοδοξία λοιπόν σε ό,τι αφορά την ε, ρευστότητα. Και η Βασιλεία το καλύπτει αυτό, γιατί η αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ζητά 20% στήριξη της ρευστότητα. Εμείς ε, περάσαμε στο 100% της κάλυψης έλλειψης ρευστότητα. Επίσης, δεν καλύπτει ακόμη πρόσβαση των ζημιών. Στις στις διαδικασίες ευεργειότητας θα πρέπει τα συστήματα εγγύηση καταθέσεων να κάνουμε σε έξι χρόνια να, να, να αποπληρώσουν την αναχρηματοδότηση. Επίσης, εξετάζουμε την ανάλυση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρούμε ότι σε, στο 90% των περιπτώσεων εξασφαλίζεται κάτι τέτοιο, ίσως και σε περισσότερες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάλυση Ευρωπαϊκή Επιτροπής, θα ήθελα να την ευχαριστήσω επ' ευκαιρία για τη συνεργασία που είχαμε και για το γεγονός ότι ε, υπέβαλε αυτή τη συμπληρωματική ανάλυση στι αρχές Οκτωβρίου, γιατί έτσι μας βοήθησε να σημειώσουμε πρόοδο. Αρχικά είχαμε κολλήσει σε μια συζήτηση για την έλλειψη μελέτη ε, επιπτώσεων, μελέτη αντικτύπου. Γιατί πρόοδος ήταν δύσκολη για πολλούς, αλλά χάρη σε αυτή την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, έχουμε διαλευκάνει αρκετά το ζήτημα. Τώρα, ένα πλεονέκτημα αυτής της πρώτης φάσης επικεντρώνεται σε φιλόδοξη στήριξη της ρευστότητα. Γι' αυτό και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρόνο για να έχουμε μείωση του κινδύνου ε, όσο έχουμε το σύστημα ώστε να μην έχουμε την ε, συζήτηση για την μείωση του κινδύνου πριν την έναρξη. Ε, γιατί κάτι θα μας εμποδίσει να ξεκινήσουμε. Θα μπορέσουμε όμως να έχουμε τη συζήτηση για περαιτέρω μείωση κινδύνου όταν ήδη θα έχουμε θεσπίσει το σύστημα που ε, αντιμετωπίζει τα, τις εύλογες ανησυχίες ε, ρευστότητας που έχουν πολλοί πολίτες. Το σύστημα εξασφαλίζει εθνικά συστήματα εγγύησεων, αντί να στηρίζει με μονομένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η χρηματοδότηση κατανέμεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν καλύπτει το 0,8% των καλυμμένων καταθέσεων. Ε, το μοιράζουμε στα 0,4% στα εθνικά DGS και 0,4% στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Σε ό,τι αφορά τον ηθικό κίνδυνο, και έρχομαι εδώ στη δεύτερη φάση, θα γίνει συζήτηση για τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν πριν περάσουμε στη φάση της ασφάλισης. Στη φάση ασφάλισης θα υπάρξει κάλυψη των υπερβολικών ζημιών. Θα πρέπει όμως να δούμε τη σειρά που σε περίπτωση ε, έχουμε σύμβαν payout ε, θα ε, καλούνται οι δανειστές να ικανοποιηθούν. Φυσικά πρώτα θα πρέπει ε, να, να προσέχουμε στο εθνικό DGS, το πρώτο 0,4%, μετά περνάμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο και σε αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο πρώτα έχουμε χρήση του μεμονωμένου υποταμείου και μετά του ε, κοινού ταμείου DIF, της, ε, κοινής, του Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων και μετά τα υπόλοιπα ε, ταμεία. Αυτό δεν συγκρίνεται με αυτό που έχουμε στο SRF, στο ενίο Ταμείο Εξήγηση Τραπεζών, αλλά είναι θέμα σειράς ατάξεις, ε, με την οποία θα καλούνται τα διάφορα τμήματα του Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων, του DIF. Τώρα, η πληρωμή, αν υπάρχουν χρήματα ή αν δεν υπάρχει αρκετή ρευστότητα από τα κράτη-μέλη, θα γίνει σε αντίστροφη σειρά σε σχέση με αυτή που σας περιέγραψα πριν από λίγο. Τέλος, και για περισσότερες λεπτομέρειες στις, σας παραπέμπω στη συζήτηση επί της εκθέσεως, θα ήθελα να τελειώσω με την ανάλυση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανάλυση των στοιχείων. Αν επιλέξετε μια τέτοια σειρά και δομή με συγκεκριμένη σειρά, στην περίπτωση που έχουμε ένα τέτοιο συμβάν, αυτό δεν περιορίζει το το σύστημα, γιατί η ελκυστικότητα ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κονδυλίου είναι ότι ενισχύεται η ισχύ του σε σχέση με τα επιμέρους εθνικά ταμεία. Χρησιμοποιώντας όμως, χρησιμοποιώντας όμως αυτή τη διτή προσέγγιση με εθνικά DGS που θα εξακολουθούν να ισχύουν όχι ως paybox απλό, κάτι που βοηθά τη συζήτηση στα κράτη-μέλη που έχουν λειτουργικά συστήματα DGS και IPS με εναλλακτικά μέτρα και μάλιστα πολύ πρό, πρόημα μέτρα παρέμβασης. Αυτά θα πρέπει να τα, μπορούν να τα συνεχίσουν γιατί είναι λειτουργικά. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτή τη διτή προσέγγιση κάτι που είναι θετικό, δεν εμποδίζουμε την ισχύ του συστήματος ισχύ γιατί μπορεί κανείς ε, να να φτάσει στο πλήρες Ταμείο Ασφάλειας Καταθέσεων αρκεί να, να κρατήσει τη σειρά προτεραιότητας που θα πρέπει να γίνει και με τον οποίο γίνεται οι ε, πληρωμές. Και μάλιστα σας παραπέμπω στη γραφική παράσταση στη σελίδα 77 με την ε, ε, ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει πόσο συγκρίσιμες είναι η... πόσο συγκρίσιμη είναι η ισχύ αυτού του ταμείου και μάλιστα υπάρχει σχεδόν απόλυτη συγκρισιμότητα. Προσπάθησα στις ε, προτάσεις μου να λάβω υπόψη τις ε, δικές σας παρατηρήσεις. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά απόψεων, όπως σας είπα, μεταξύ των ομάδων και εντός των ομάδων. Η συζήτηση ε, δεν θα, στην αρχή δηλητηριάστηκε από την αιρεσιμότητα. Δεν θα πρέπει ε, να αποτελματοθούμε σε αυτό το σημείο και προ, περιορίζοντας στο δεύτερο σημείο Μα δίνει την πολυτέλεια του χρόνου για να έχουμε περαιτέρω συζήτηση για την αιρεσιμότητα. Επίση λαμβάνουμε υπόψη ε, τι των χωρών που έχουν τέτοια συστήματα εγγύησεων και μάλιστα λειτουργικά. Και επίση λαμβάνουμε υπόψη την εύλογη ανησυχία των πολιτών στα κράτη-μέλη που λένε ότι εγώ δεν εμπιστεύομαι το εθνικό σύστημα εγγύησεων. Δεν θεωρώ ότι μέσα σε μία εβδομάδα, αν ε, δημιουργηθεί κρίση, θα μπορέσει να πληρώσει το σύστημα. Και αυτό και προβλέπεται η αύξηση της στήριξης ρευστότητας. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το θέμα και περιμένω τις απόψεις των συναδέλφων. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε πολύ συχνά την ευκαιρία και στο μέλλον να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή και περιμένω τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Εστέρ. Ξεκινάει τώρα η συζήτηση με τους κοιόδης συζητητές. Ο κύριος ε, Φερνάντες πρώτος. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Την ε, μελετήσαμε εμπεριστατωμένα τις τελευταίες μέρες και πιστεύω ότι θα αποτελέσει το μύτο της Αριάδρης για τη συζήτηση και στο μέλλον. Είναι σημαντικό, όπως είπε και η Έστερ Ντελάνγκε, χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραμείνει ζωντανός ο κανονισμός και η έκθεση. Και ίσως ο καλύτερος τρόπος είναι να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις για να τον κρατήσουμε ζωντανό και να καταλήξουμε και στη συμφωνία. Τώρα, ας ε, σας υπενθυμίσω γιατί συζητούμε αυτό το το σύστημα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύης των Καταθέσεων. Η κρίση στην Ευρωζώνη μεταξύ 2010 και 2012 σχεδόν ε, διέλυσε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ήταν μεγάλη κραδασμή και το, τον Ιούνιο του 2012 το Συμβούλιο αποφάσισε να θεσπίσει την Τραπεζική Ένωση με διπλό στόχο. Ο πρώτος στόχος ήταν να ελαχιστοποιηθούν οι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι εντός της Ευρωζώνης και ο δεύτερος στόχος να δι, ο κίνδυνος μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ε, ε, ιδρυμάτων και των Εθνικών Κορβανάδων. Και αυτοί αυτή η οδήγησαν στο μηχανισμό, τον ενιαίο μηχανισμό, το Ταμείο Εξυγίασης και το Μηχανισμό Εξυγίασης και τώρα έχουμε τη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων. Θέλουμε να μειώσουμε τους κινδύνους του τραπεζικού συστήματος και ένας τρόπος για να μειώσουμε τους κινδύνους αυτούς είναι ε, τον κίνδυνο, τον δεσμό μεταξύ τραπεζών και κρατών. Οπότε Υπό αυτό το πρίσμα μπορούμε να ερμηνεύσουμε την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύης Καταθέσεων με βάση αυτά τα κριτήρια. Τα προβλήματα της Ευρωζώνης δεν δημιουργήθηκαν βέβαια από το δημόσιο χρέος που θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει τραπεζικές κρίσεις. Το αντίθετο, οι τραπεζικές κρίσεις ε, εξαιτία του ατελού σχεδιασμού της Ευρωζώνης προκάλεσε τις δημοσιονομικές κρίσεις. Πάντως η πρόταση της κυρίας ε, Ντελάγκε, κατά τη γνώμη μου, ε, περιέχει και σημαντικά προβλήματα. Γιατί δεν ανταποκρίνεται στο στόχο της ελαχιστοποίησης των κινδύνων. Ούτε απομονώνει τα κράτη από και τους εθνικούς κορβανάδες από τις τραπεζικές κρίσεις. Το σύστημα που προτείνει η κυρία Ντελάγκε με, μέσα σε μία επταετία, όχι, η πενταετία από το 2019, με, με μία εξασφάλιση της ρευστότητας ε, και μία αιρεσιμότητα που μερικές φορές είναι πολύ περιοριστική. Γιατί αν παραμείνουν αυτές οι προϋποθέσεις, ουδέποτε θα περάσουμε στη δεύτερη φάση του συστήματος που προτείνει η συγγετρία. Πάντως ακόμη και αν συντρέξουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις θα φτάσουμε σε ένα σύστημα ότι ακόμη το 50% των ζημιών θα καλύπτονται από τις εθνικές ασφάλειες. Και ένα τμήμα θα καλυφθεί και από την εθνική ασφάλεια, ώστε αυτή η αμοιβαιοποίηση, αυτό το 0,2, αυτός ο επιμερισμός των κινδύνων, μόνο το 0,2 των εγκειμένων καταθέσεων περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Αν θέλουμε όμως να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, θα πρέπει να συζητήσουμε τι είδους προϋποθέσεις θέλουμε για να περάσουμε στη δεύτερη φάση. Επίσης θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι στη δεύτερη φάση η κίνδυνη θα είναι ακόμα μεγαλύτερη... σε ένα σύστημα με μεγαλύτερο επιμερισμό. Γιατί όσο λιγότερη με έχουμε τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο έχουμε. Αν θέλουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο λοιπόν θα πρέπει να αυξήσουμε ε, είναι μάλλον να λάβουμε υπόψη ότι όσο μεγαλύτερη αμοιβεοποίηση, όσο μεγαλύτερο επιμερισμό έχουμε, λιγότερο κίνδυνο θα αναλαμβάνουν τα μέλη του συστήματος. Δεν ξέρω ποιε πρέπει να είναι εκ των προτέρων προποθέσει, το βαθμό επιμερισμού, αν θέλουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε και να συζητήσουμε επίση πώ θα απομονώσουμε ε, τα κράτη από τι τραπεζικέ κρίσει και τους εθνικούς προϋπολογισμούς από τις τραπεζικές κρίσεις. Πάντως επαναλαμβάνω, ε, ε, η κρίση του 2012 ήταν ε, η αιτία για την, για την πρόταση της Τραπεζικής Ένωσης, αλλά η κρίση αυτή δεν έχει ακόμη όλο τερματιστεί. Γιατί σε περίπτωση απολειών ακόμη ε, οι εθνικές ασφάλειες αναλαμβάνουν το κόστος ε, των ζημιών. Γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε τους εθνικούς ε, προϋπολογισμούς. Οπότε αν μεταβούμε σε ένα σύστημα που είναι λιγότερο ασφαλές από ό,τι θα όφιλε και ε, με προβληματίζει η μέθοδος της κυρίας Δελάνκε για να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους και να έχουμε λιγότερη ελαχιστοποίηση των κινδύνων από ό,τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω, γιατί αν δεν καταφέρουμε να, να διαρρήξουμε αυτόν τον κίνδυνο μεταξύ τραπεζών και εθνικών προϋπολογισμών, τότε δεν θα καταφέρουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα που δημιούργησε η κρίση και που έδωσαν λαβή για την πρόταση της Τραπεζικής Ένωσης. Σίγουρα θα συνεχίσουμε να αγγίπτουμε σε αυτά τα θέματα και η ομάδα μου είναι πρόθυμη για περαιτέρω συζήτηση και διαλλακτική, αλλά θα πρέπει πρώτα να δούμε πώς θα ελεγχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, όχι μόνο εξάντε κινδύνους, αλλά και κινδύνους του ίδιου του τραπεζικού συστήματος και πώς θα απομονώσουμε τους εθνικούς προϋπολογισμούς από, θα τους φέρουμε στο πυρόβλητο αυτών των τραπεζικών κρίσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για το ΙΣΙΑΡΟ, κύριο Λουκέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δικαστώ τον κύριο Λούνες και πάλι, τον σκιώδη εισηγητή του ECR, ο οποίος ζητά συγγνώμη γιατί έχει άλλες υποχρεώσεις. Λοιπόν, θα διαβάσω μία δήλωσή του. Ο κύριος Λούνης ευχαριστεί την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Είναι σαφές ότι εκμεταλλεύτηκε τους προηγούμενους δύο μήνες. Η πρόταση είναι οπωσδήποτε μια σωστή αφετηρία. Ο σκιώδης μας εισηγητής πιστεύει πως όλες οι πολιτικές ομάδες εδώ πέρα θα πρέπει να δεχτούν τουλάχιστον κάποια από τα στοιχεία της έκθεσης. Όμως το ECR βλέπει κάποιες αρχές, ιδέες που οπωσδήποτε αξίζουν στήριξη, ενώ άλλες όχι. Θα ξεκινήσω με αυτό το οποίο θεωρεί σοβαρά ζητήματα και μετά θα ε, τελειώσω με κάποια θετικά σημεία. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Λούνες δεν συμφωνεί με τον χρονισμό της αιρεσιμότητας. Θα έπρεπε να είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν όροι πριν ξεκινήσει το σχέδιο. Οπότε τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων θα μπορούν να ζητήσουν χρηματοδότηση, ολόκληρη τη χρηματοδότηση που τους λείπει για να χρηματοδοτήσουν την έλλειψη ρευστότητας πριν εκπληρωθούν οι όροι. Αυτό πρέπει να αλλάξει γιατί αν είναι να ζητήσουμε από τις ευρωπαϊκές τράπεζες να διασώσουν παραδείγματο χάρη του Ιταλούς καταθέτες θα πρέπει να μπορούν να εξετάσουν ακριβώς την ασφάλεια αυτών των καταθέσεων. Αλλιώς το ίδιο κινδυνεύει να ε, μην ε, μοιράζεται τον κίνδυνο, αλλά την παρελθούσα ιστορία. Επίσης πρέπει να γίνει κάποια περισσότερη δουλειά όσον αφορά τους όρους, ειδικά κοιτώντας την έκθεση των κρατών. Ο κ. Λούνας εκτιμά αυτά τα οποία αναφέρονται στην έκθεση, αλλά θεωρεί ότι η διατύπωση δεν είναι αρκετά στιβαρή. Θεωρεί ότι οποιαδήποτε αμοιβεοποίηση της προστασίας των καταθετών έχει νόημα μόνο εάν αντιμετωπιστεί το ζήτημα του κινδύνου των διαφόρων κρατών. Επίσης, το ζήτημα του εάν τα ζητήματα αυτά είναι επαρκώς ασφαλή για το ΙΔΙΣ και αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το πολιτικό. Δεν μπορεί να το αφήσουμε στην Κομισιόν. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να έχουν λόγο εδώ. Τρίτον, ο σκιώδης του ΙΣΙΑΡ θα ήθελε να επαναλάβει πως οι δυνατότητες για να επιτευχθεί μια ανάκαμψη από τις ε, διαδικασίες χρεοκοπίας είναι κάτι το δύσκολο το οποίο μπορεί να γίνει μέσω του εθνικού νομοθετικού συστήματος, γι' αυτό δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί θα πρέπει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ε, κάλυψης ε, των ασφάλισης των καταθέσεων να καλύπτει αυτές τις απολύες. Κατόπιν, ακόμα και αν έχουν μειωθεί επαρκώς οι κίνδυνοι, τότε ο κύριος Λούνες ε, θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Ταμείο να σπάσει σε δύο μέρη. Είναι μια πολύ καλή λύση την οποία προτείνει η συγγήτρια. Δηλαδή πρώτα αναλαμβάνει κανείς ευθύνε του και μετά έχει ε, την αλληλεγγύη βεβαίως. Και βεβαίως αυτό θα, θα υπάρχει και για το κοινό ταμείο το οποίο θα βασίζεται στον κίνδυνο. Επίσης υπάρχουν τα ζητήματα αυτά του χρονισμού και της αιρεσιμότητας, τα οποία αν επιληθούν τότε η λειτουργία του Ταμείου, όπως προτείνει η συγγήτρια, ίσως αποτελέσει μια βάση για μελλοντικές συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε Έστερ για πολλή δουλειά που κάνετε εδώ είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα και οι σημερινές συνθήκες ε, πέρασε ένας χρόνος μετά από την πρόταση της Κομισιόν δουλέψαμε σκληρά, αναμέναμε την εκτίμηση αντικτύπου και ήθελα να ξεκινήσω με δύο παρατηρήσεις πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό κατά την απόψή μου να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση και αυτό που εκτιμώ Ιδιαίτερα είναι ότι προσπαθεί να βρει μια οδό η έκθεση αυτή για να προχωρήσουμε. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ένα κοινό συμφέρον, την η χρηματοοικονομική σταθερότητα. Και χωρίς να θέλω να αναφέρω την επικαιρότητα, μπαίνουμε σε έναν νέο κόσμο, πιστεύω, όπου οι εξωτερικές πηγές αποσταθεροποίησης ε, ε υπάρχει κίνδυνος να θέσουν διπλωματικά προβλήματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να διατηρήσουμε ένα κοινό ορίζοντα, ένα κοινό στόχο. Συνεπώ η συζήτηση έχει αλλάξει πορεία. Ε, ε, είναι πολύ εθνική πλέον η συζήτηση και ε, εθνικοποιούμε ζητήματα τα οποία είναι κοινά όμως για όλους όπως η προστασία των αποταμιευτών. Δεν καταλαβαίνω γιατί ορισμένε χώρες πρέπει να ισχυρίζονται ότι η θέλησή τους να προστατεύσουν τους ε, αποταμιευτές είναι ισχυρότερη από άλλες. Ε, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κοινό σύστημα στο οποίο έχουν εμπιστοσύνη όσοι αποταμιεύουν. Υπό αυτό το πνεύμα θα ε, εργαστούμε. Η πρόταση της Αστέρα αλλάζει πολλά από αυτά που προτείνει η Κομισιόν. Δεν θα τα αναλύσουμε σήμερα, αλλά θα τα συζητήσουμε και με τους συναδέλφους της ομάδας. Όπως είπε και η συγγήτρια, υπάρχουν διχογνωμίες μεταξύ ομάδων αλλά και εντός των ομάδων. Απλά σήμερα δίνω εγώ μια πρώτη αντίδραση για πέντε σημεία. Το πρώτο. Υπάρχει μια αλλαγή αρκετά σημαντική σε σχέση με αυτά που προτείνει η Κομισιόν. Και στην παρούσα φάση δεν ξέρω τι να σκεφτώ ειλικρινά. Αρχικά η Κομισιόν ε, σκεφτόταν ένα σύστημα που θα τροφοδοτούν οι τράπεζε και εδώ έχουμε ένα ε, σύστημα το οποίο βασίζεται στα DG. συστήματα. Ε, οπότε εκεί πρέπει να δούμε κάπως τη τεχνική πτυχή των πραγμάτων. Δεύτερη παρατήρηση όσον αφορά τη λειτουργία του α, Ταμείου Εγγύησης. Θα παρέχει ρευστότητα, θα απορροφά τις ε, ζημίες, ε, θα χρησιμοποιεί αμοιβαιότητα. Ε, αυτό προτείνει η συγκήτρια γιατί όχι, ναι, συμφωνώ με το να επιμείνουμε στη ρευστότητα και στην δυνατότητα ταχείας αντίδρασης. Διότι ουσιαστικά σκοπός αυτής της νομοθεσίας είναι να αποφύγουμε τραπεζικό πανικό και ε, ανεξέλεγκτες κινήσεις χρημάτων και ο κόσμος να υποφελείται από εγγυήσεις που θα θεσπίζονται από ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης θεωρώ ότι είναι θετικό που δεν υπάρχει ε, διαμερισματοποίηση στο πλαίσιο διότι όλα αυτά εισάγονται εντός μιας ευρωζώνης ε, οπότε κάποιες διασυνοριακές τράπεζες μεγάλοι όμιλοι τη Ευρωζώνη ουσιαστικά δραστηριοποιούνται διασυνοριακά. Οπότε όλα αυτά θα χρειαστούν κάποια ανάλυση. Ομολογώ ότι η διαφορά μεταξύ τη αμοιβαιοποίηση και τη επανασφάλιση είναι κάτι που πρέπει να το ξαναδούμε. Πέρασα τη νύχτα στο CNN, οπότε συγχωρέστε με αν δεν τα λέω καθαρά. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε και πολιτικά και οικονομικά, εννοείται. Εδώ έρχομαι στο τρίτο μου σημείο, στην αιρεσιμότητα. Προσωπικά, θα ήθελα να το ξαναπώ, η Άλντε δεν είναι κατά τη αιρεσιμότητα. Αντιθέτω, απλά πρέπει να γίνει σοβαρά. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη. Προσωπικά, ναι, καθεν πίστευα ότι χρειάζονταν προϋποθέσεις, ε, κάποια αιρεσιμότητα για αυτή το quality review, να δούμε κατά πόσο υπάρχει ένα σύστημα εποπτεία το οποίο ενδεχομένως χρήζει αναθεώρηση. Ε, για να γίνει πιο αποτελεσματικό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με όλα αυτά, αλλά πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο έχουμε την αιρεσιμότητα και ποιο είναι ο βαθμό αιρεσιμότητα. Πρόκειται για μια παράλληλη δουλειά που γίνεται παράλληλα με άλλα ζητήματα ή πρόκειται για μια δικλίδα ασφαλείας. Οπότε θέλω να διαφοροποιήσουμε κάπως τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις ισχύω και τις συνθήκες εισόδου. Και κάτι που με φοβίζει είναι η θέση ισχύ ενό ευρωπαϊκού πλαισίου για τη χρεοκοπία των επιχειρήσεων. Είμαι υπέρ του να υπάρχει τέτοιο πλαίσιο και μάλιστα πιστεύω ότι ο Επίτροπος Ντομπρόφσκης έχει αναφερθεί σε αυτό στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών με όλα τα ζητήματα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό. Απλά λέω ότι τελικά μπορεί να δημιουργήσουμε μια δικλίδα ασφαλείας στα Υπουργεία ε, Δικαιοσύνης των χωρών μας. Ε, γιατί στα περισσότερα κράτη-μέλη τα Υπουργεία Δικαιοσύνης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Και εκεί η βασική ανησυχία θα είναι να υπερασπιστούμε το εθνικό δίκαιο περισσότερο από το να δημιουργήσουμε την Τραπεζική Ένωση. Οπότε πρέπει να το προσέξουμε λίγο αυτό. Τώρα για τη μείωση του κινδύνου, το risk reduction που είναι το πιο πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα, δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ιδέα του να κινηθούμε προς την κατεύθυνση μιας μείωσης ε, ε, τις ε, τάσεις ε, χρέωσης των κρατών της Ευρωζώνης. Αυτό που μου δημιουργεί κάποια ερωτηματικά είναι ότι είναι αυτή η καλύτερη οδός ή μήπως αυτή τη στιγμή εμένουμε στο να εξετάζουμε ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να είχε λύσει το six-pack και όπου η Κομισιόν θα έπρεπε να είχε αναλάβει περισσότερες ευθύνη κατά την απόψή μου από ό,τι κάνει αυτή τη στιγμή και για ορισμένες χώρες και αυτές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες αν καταλαβαίνετε αυτό που θέλω να πω δηλαδή με την αιρεσιμότητα. Υπάρχει κάποια αιτιολόγηση όσον αφορά το σύνδεση μεταξύ ε, εθνικού ε, χρέους ε, και δημοσίου χρέους. Λοιπόν, γρήγορα τα δύο τελευταία σημεία αναφέρθηκε επίσης και από τον κύριο Λούκε. Υπάρχει το ζήτημα του legacy. Ό,τι και να κάνουμε για το μέλλον, ακόμα και αν βελτιώσουμε τις περιπτώσεις χρεοκοπίας και όλα αυτά, θα έχουμε πίσω μας κάτι που έχει ήδη γίνει. Η κατάσταση των τραπεζών δεν πρόκειται να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Το στόκ αυτό θα υπάρχει στις τράπεζες. Δεν υπάρχει απλή λύση. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και τελευταίο, εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό το ότι απομακρύνουμε την διακυβερνητική συμφωνία και κάτι τέτοιο ενδεχόμενο το είχαμε δει στην προηγούμενη θητεία με την Ελίζα Φερέρα τι είχε γίνει. Είχε ε, στερηθεί τότε το Ευρωκοινοβούλιο αρμοδιότητες για θέματα εσωτερική αγοράς τις οποίες έπρεπε να έχει. Οπότε το θέμα είναι να μην υπερασπιστούμε τα δικά μας δικαιώματα. Είναι, πρέπει να φτιάχνουμε τις νομοθεσίες με το σωστό τρόπο, με την συναπόφαση και με τον ε, ρόλο των υπουργών να υπάρχει. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Ευχαριστούμε πολύ συνεχίζουμε, θα είμαστε επικοδομητικοί ώστε να προχωρήσουμε. Αλλά για άλλη μια φορά, όπως είπε και η συγγήτρια, δεν πρέπει η αιρεσιμότητα ή οι συζητήσεις να καταλήξουν στην αναζήτηση αιτιολογιών για απραξία τελικά. Είναι κάτι το οποίο κατά εμάς είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Τραπεζικών Καταθέσεων αποτελεί τον τρίτο πυλώνα ενός σχεδίου για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μια διαδικασία την οποία έχει χαιρετήσει και εγκρίνει με ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάρτιο του 2016. Και ήδη καθυστερεί αυτή η διαδικασία. Θεωρώ επικίνδυνη κάθε περαιτέρω καθυστέρηση ή αποδυνάμωση αυτής της δρομολογημένης τραπεζικής ενοποίησης. Επικίνδυνη και για τους Ευρωπαίους πολίτες, για τους Ευρωπαίους καταθέτες, για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και θέλω να πω και πιο καθαρά αυτό που υπενήχθηκαν κάποιοι από τους προηγούμενους ομιλητές. Θεωρώ ότι η εκλογή Τραμπ προσθέτει αβεβαιότητα, αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία, ανησυχίες και το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την ώρα είναι να συνεχίσουμε να αναβάλουμε, να καθυστερούμε και να βλέπουμε το θέμα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ενοποίησης μέσα από τα χρωματιστά γυαλιά της σκοπιμότητας εθνικών εγωισμών ή στενά τραπεζικών ή συντεχνιακών συμφερόντων. Σε ό,τι αφορά την έκθεση της ε, κυρίας Δελάνγκε. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω ε, για την έκθεση που μας έστειλε στις 3 Νοεμβρίου. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στη σημαντική καθυστέρηση της υποβολής αυτής της έκθεσης, περίπου 20 μέρες, σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχαμε συμφωνήσει, που μας περιορίζει το χρόνο για μια ουσιαστική συζήτηση και κατάθεση τροπολογιών και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε αναγκαστικά τον επανακαθορισμό του χρονοδιαγράμματός μας εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης στην κατάθεση της αναφοράς της εισηγήτριας. Θεωρώ επίσης σημαντικό μέσα από το διάλογο μεταξύ μας να βρούμε εκείνο το πλαίσιο που σε συμφωνία και με το ψήφισμα που έχουμε ήδη εγκρίνει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάρτιο που μας πέρασε, να εξασφαλίσει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης καταθέσεων αποτελεσματικού και εντός των χρονικών πλαισίων που έχουν προταθεί από την Επιτροπή. Θεωρώ ότι οκτώ χρόνια είναι υπεραρκετά για να εξασφαλίσουμε τα αναγκαία βήματα. Δημιουργώντας και όχι υποσκάπτοντας και υπονομεύοντας τη δημιουργία του τρίτου πυλώνα το ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει δεν είναι αν πρέπει να δημιουργηθεί το έντις στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής ή πότε θα είναι οι κατάλληλες συνθήκες, αλλά να εργαστούμε με την ευρύτερη δυνατή συνένεση μεταξύ μας, ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό έντις που βήμα-βήμα μέσα στα επόμενα 8 χρόνια θα διασφαλίζει και τους καταθέτες σε όλες τις χώρες μέλη και θα ενισχύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Διαφορετικά θα περάσουμε το μήνυμα ότι το Ευρωκοινοβούλιο λέει ναι αλλά κάρτ στην ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος, ναι στον πρώτο πυλώνα, ναι στον δεύτερο πυλώνα, αλλά να το σκεφτούμε, μάλλον, ίσως, όχι, θα δούμε, Ας καθυστερήσουμε μερικά χρόνια ή ας το ψαλιδίσουμε όταν ερχόμαστε στον τρίτο πυλώνα που είναι ο πιο σημαντικός για τους Ευρωπαίους πολίτες, για τους Ευρωπαίους κατα... καταθέτες. Αυτό το λάθος μήνυμα δεν νομίζω ότι πρέπει να το στείλουμε. Η αναφορά της ε, κυρίας Δελάγκε ουσιαστικά διαιωνίζει την υπάρχουσα ανισορροπία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους τρεις πυλώνες, αφήνοντας τους καταθέτες να έχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας και εμπιστοσύνης, ενεργώντας έτσι αποτρεπτικά στη δημιουργία των συνθήκων για την ολοκλήρωση των σταδίων του έντις. Θα συμφωνήσω ότι το περιεχόμενο, content, η χρονική στιγμή, timing και η αιρεσιμότητα, conditionality, είναι πολύ σημαντικά και αλληλένδετα στοιχεία. Το ερώτημα είναι όμως πώς τα προσεγγίζουμε. Και δεν συμφωνώ καθόλου να βαφτίζουμε την πρόταση της Επιτροπής, μαξιμαλιστική ή φιλόδοξη, αντί να συζητούμε το πώς θα εφαρμοστεί μέχρι το 2024 όπως προτείνεται. Η αναφορά δεν είναι επίσης συνεπής και με τους άλλες πυλώνες της τραπεζικής ενοποίησης αφού δεν συνδέει την προστασία του καταθέτη και τον έλεγχο των κυρίων παραγόντων που επηρεάζουν τον κίνδυνο των καταθετών. Η αναφορά επίσης τίνει να διαιωνίζει τα διαφορετικά χρηματοπιστωτικά backstops με αποτέλεσμα τον κατακαιρματισμό της τραπεζικής αγοράς, αφού το κριτήριο της βάσης τοποθεσίας της τράπεζας παραμένει έτσι καθοριστικό. Ως αποτέλεσμα, κινείται αντίθετα στις αρχές της μείωσης της ηθικής ζημιάς, moral hazard, και της εθνικής μη διάκρισης national indiscrimination. Επίσης μειώνοντας τους πόρους του ίδις που διατίθεται συνολικά στο 0,4 από 0,8 που προτείνει η Επιτροπή, δηλαδή 50% μείωση για την κάλυψη καταθέσεων, ουσιαστικά μειώνει τον έλεγχο και την διασπορά του κινδύνου. Το σύστημα αυτό δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τόσο αποτελεσματικά όσο ένα ολοκληρωμένο έντις την εξάπλωση μιας διασυνοριακής τραπεζικής κρίσης. Η μη ξεκάθαρη πρόταση επίσης για το δανεισμό του έντις από την αγορά σαν τελευταία λύση, η οποία θα αποπληρώνεται από τον εμπλεκόμενο εθνικό DGS, μαζί με την κατάργηση των έκτακτων εισφορών, μειώνει δραστικά και την δυνατότητα απορρόφησης των ζημιών από το Ταμείο. Καταπατάται έτσι η αρχή της ουδετερότητας κόστους και της αποτελεσματικότητας cost neutrality and efficiency, με την ουσιαστική παράταση της σύνδεσης κράτους τραπεζών. Η προτινόμενη αναφορά από την κυρία Ντελάνγκη επίσης ενισχύει την γραφειοκρατία αναφορικά με τις συμφωνίες που απαιτούνται για την υπογραφή δανείων, όπως επίσης και τη δημιουργία αριθμού υποταμείων, sub-funds, με βάση το διαφορετικό επίπεδο κινδύνου. Επίσης τίθενται νομικά θέματα σχετικά με την επιβολή υποχρέωσης σε ένα εθνικό... Νομίζω ότι συζητάμε μεγάλη καθυστέρηση ένα σοβαρό θέμα και δεν έχω... Ε, δεν είχαμε βάλει κάποιο όριο, κύριε Πρόεδρε. Επίσης τίθενται νομικά θέματα σχετικά με την επιβολή υποχρέωσης σε ένα εθνικό DGS να λάβει δάνειο με προϋποθέσεις που ορίζονται από ένα τρίτο μέρος. Είναι προφανές επίσης ότι είμαστε αντίθετοι στην πρόταση για δύο φάσεις, όπως αυτές προτείνονται, ουσιαστικά βάζοντας ερωτηματικά για την αναγκαιότητα και την δυνατότητα της ύπαρξης του σταδίου της πλήρους ασφαλείας, full insurance. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζω ότι καλωσόρισε το Μάρτιο του 2016 την πρόταση της Επιτροπής και τη διαδικασία των τριών σταδίων με την σταδιακή μεταφορά από το reinsurance στο full insurance, όπως και μια παράλληλη πορεία του επιμερισμού του κινδύνου με την μείωση του κινδύνου, κάτι που επιμελώς αποσιωπάται στο σχετικό επεξηγηματικό κείμενο. Λυπάμαι, αλλά κατά την άποψή μας η έκθεση της κυρίας Δελάνγκη κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, αφαιρώντας σημαντικά θετικά στοιχεία από την πρόταση της Επιτροπής και εμπεριέχει και αρκετά προβληματικά στοιχεία για τα οποία θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Θα ήθελα πριν κλείσω να προτείνω να καλέσουμε στην Επιτροπή μας την Κομισιόν για να μας παρουσιάσει αναλυτικά την ανάλυση που δημοσίευσε τον Οκτώβριο όσο και για να συζητήσουμε και με την Κομισιόν τις σημαντικές διαφορές και αποκλήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην πρόταση της Κομισιόν και στην πρόταση της κυρίας Ντελάγκε. Συμπερασματικά, η προτινόμενη αναφορά της ε, συναδέλφου Ντελάγκε θέτει κατά τη γνώμη μου σε κίνδυνο μια υγιή και εναρμονισμένη τραπεζική ενοποίηση, δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα και καθυστερήσεις και ουσιαστικά διαιωνίζει τον κατακαιρματισμό της τραπεζικής αγοράς και την μη ουσιαστική προστασία των ευρωπαϊκών καταθετών. Αντικατοπτρίζει μια πολιτική που θέλει την Τραπεζική Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση la carte και που στηρίζει την ευάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο όπου συγκεκριμένα εθνικά, τραπεζικά ή συντεχνιακά συμφέροντα εξυπηρετούνται. Και με αυτή την carte προσέγγιση που τη θεωρώ πολύ εγωιστική, λογικό είναι να μην συμφωνούμε καθόλου. Ευχαριστώ. Thank you για το θέμα του χρονοδιαγράμματος, ε, του χρονικού σημείου που αναφέρατε, το συζήτησα με την εισηγήτρια και συμφωνήσαμε ε, να παρατείνουμε ελαφρώς την προθεσμία για τις 16 Δεκεμβρίου για να έχουν οι σκιώδεις σε επαρκή χρόνο να μελετήσουν αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ο Φίλιπ Λάμπερτς είναι επόμενος ομιλητής. Καλημέρα Ευρώπη. Α, συγγνώμη δεν είναι συνήθις τρόπος έναρξη μιας ομιλίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εστέρ για το έργο της, γιατί πραγματικά ε, σου δίνω τα εύσχημα που δεν θέλεις ε, να αναπαγείς αυτή η προσπάθεια, αλλά να δοθεί μία πνοή. Και οι προαλήσαντες είπαν ότι συμμερίζονται αυτό το στόχο, να υλοποιήσουμε κάτι και μάλιστα κάτι σημαντικό κάποιοι και μάλιστα συγκεκριμένα ο κύριος Λούκε που παρέθεσε τη γνώμη του κυρίου Λούνς διευκρίνησε ότι δεν θέλει πρόοδο, δεν επιζητεί πρόοδο. Οπότε, Εστέρ, το πρώτο πράγμα που θα σου θα σε παρακαλούσα να κάνεις είναι να διαλέξεις την πλειοψηφία που θα ήθελες, γιατί δεν είμαι βετεράνος ευρωβουλευτής, αλλά είμαι αρκετά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να γνωρίζω ότι δεν είναι καλή ιδέα να εξοδέψουμε πολιτικό κεφάλαιο και να κάνουμε υποχωρήσεις σε ανθρώπους που σε τελική ανάλυση δεν θα υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Οπότε διάλεξε τους συμμάχους σου και την πλειοψηφία αν θέλεις να υλοποιήσεις κάτι. Και μην χάνεις τον χρόνο σου με ανθρώπους που πραγματικά ε, επιζητούν την αποτυχία αυτού του σχεδίου. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να βρούμε την ε, σωστή ισορροπία για το χρονικό σημείο, το περιεχόμενο και την αιρεσιμότητα, αλλά όπως είπαν και κάποιοι προλαλήσαντες, θα πρέπει να είναι σαφές επίσης ότι εδώ δεν μιλούμε για κάτι απλώς προαιρετικό. Ε, δεν είναι κάτι που ε, θέλουμε να κάνουμε για να σώσουμε το ενιαίο νόμισμα που χρειαζόμαστε μια πλήρη τραπεζική ένωση. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, αλλά όχι επαρκής όρος. Βέβαια, μερικοί είναι πολύ συγκαταβατικοί και λένε «Ε, εντάξει, επιβίωσε ούτως ή άλλως η Ευρωζώνη, η κρίση περνάει, είμαστε σχετικά ασφαλείς, ε, ε, μπορούμε να συνεχίσουμε. Όχι, όχι. Δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε, γιατί αν δεν ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση και πολλά άλλα θέματα, δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης για παράδειγμα, αλλά εδώ μιλούμε για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, το ίδιο το ευρώ θα διακυβευτεί και θα διατρέξει κίνδυνο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αίσθηση ε, της ε, επίγουσας ανάγκης. Και σίγουρα οι προτάσεις δεν είναι επαρκείς ε, και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιμέρους ευαισθησίες. Πάντως είναι σαφές ότι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω μας πορεία. Ίσως ε, δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για την ερμηνεία που έδωσες στη μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ, όπως διαβάζω, ε, λέω, ε, λέω ότι όσο περισσότερη αμοιβαιοποίηση και διαφοροποίηση υπάρχει, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα οικονομικά ωφέλη, τα νομισματικά ωφέλη. Και δεν είναι όλες οι προτάσεις εξίσου επωφελείς και σταθεροποιητικές. Εγώ διαφορετικά ερμηνεύω λοιπόν αυτή τη μελέτη επιπτώσεων. Και όπως ε, σου απάντησα χθε στο mail, θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα οι σκιώδεις ηγητές να συνεργαστούν με την εισηγήτρια και να συνομιλούσουμε με τους συντάκτες της ε, μελέτης επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να έχουμε μια κοινή ερμηνεία αυτής της μελέτης αντικτύπου. Τώρα για τις δύο φάσεις. Πέραν της κάλυψης ε, της έλλειψης ρευστότητας, συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μία ε, περαιτέρω, με, με έναν το όριο κάλυψης ε, των επιπλέον ζημιών θα πρέπει να καλυφθεί στη φάση 1. Τώρα θα πρέπει να δούμε πού θα πρέπει να είναι αυτό το ανώτατο όριο. Ίσως το 40% είναι το ανώτατο όριο της κάλυψης. Αλλά κάτι τέτοιο ήδη θα πρέπει να εμφανίζεται ήδη από την πρώτη φάση. Τώρα για τη δεύτερη φάση, όπως προτείνεις, ε, συμφωνούμε ότι η πρόταση είναι κατάλληλη για όλες τις τράπεζες που βρίσκονται κάτω από το κατόφλι του ενιαίου υποπτικού μηχανισμού. Ε, δηλαδή ισχύει για τις μη συστημικές τράπεζες αυτό που προτείνει. Αν όμως μιλάμε για τράπεζες που πληρούν τα κριτήρια του SSM, του ενιαίου υποπτικού μηχανισμού, τότε εκεί θα χρειαζόμαστε ένα πλήρες σύστημα αντασφάλισης και πλήρη κάλυψη ζημιών και όχι μόνο κάλυψη του, των, επιπλέον, ε, υπερβολικών ζημιών. Και αν έχουμε μια τοπική πυρκαγιά, αρκεί το τοπικό πυροσβεστικό σώμα. Αν είναι όμως εξαπλωμένη η πυρκαγιά, σε όλη την πόλη για παράδειγμα, θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια από τις γειτονικέ πόλεις και από τα δικά τους πυροσβεστικά σώματα για να α, ελέγξουμε την πυρκαγιά. Οπότε χρειαζόμαστε ένα πλήρες σύστημα αντασφάλισης. Συμφωνώ με την ιδέα του, της μείωσης του κινδύνου και ήμασταν στεναροί σε αυτό το σημείο. Βέβαια εδώ ακούω δύο διαφορετικά θέματα, δύο διαφορετικούς, ε, δύο διαφορετικές μελωδίες. Οι, μεν ε, ανησυχούν για τις ευπάθειες του συστήματος που δεν αντιμετωπίστηκαν και εδώ θα έλεγα στους Γερμανούς συναδέλφους ότι δεν είναι τα αδύναμα ε, συστήματα του Νότου μόνο, ενώ έχουμε ένα από τη μια και το ισχυρό γερμανικό σύστημα από την άλλη. Νομίζω ότι η πιο το πιο επικίνδυνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι η Deutsche Bank. Και αν ξέρω σωστά γερμανικά, το Deutsche, από το Deutsche Bank σημαίνει γερμανική τράπεζα. Και είναι η πιο επικίνδυνη τράπεζα. Δεν είναι μοναδική. Αλλά θα συμβούλευα αυτούς που βλέπουν κάπως ε, υποτιμητικά κάποια άλλα συστήματα τραπεζικά σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, να συμμαζέψουν και να διορθώσουν τα του οίκου τους πρώτα πριν ε, κοιτάνε υποτιμητικά τους υπόλοιπους. Έχουμε λοιπόν ε, αυτού αυτούς που λένε ότι θα πρέπει να διορθώσουμε τα προβλήματα, αλλά υπάρχουν και άλλοι που λένε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σύνθημα της μείωσης κινδύνου πρόσχημα για αδράνεια γιατί τελικά στόχος τους είναι να μην μειωθεί ο κίνδυνος. Εγώ λοιπόν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι αν αμοιβοποιήσουμε τον κίνδυνο και αυτό είναι απαραίτητο και αναφυσβήτητο, τότε θα πρέπει ταυτόχρονα να τον μειώσουμε αυτόν τον κίνδυνο. CRD, BRD, όλα αυτά που κάναμε ε, δεν αρκούν. Η επάρκεια κεφαλαίων, η, η εξυγίαση δεν αρκούν. 6, 7, 8 χρόνια από την έναρξη της κρίσης Έχουμε ακόμη ορολογιακές ε, βόμβες ε, ε, τύπου Deutsche Bank ή τύπου κάποιων Ιταλικών τραπεζών και όλα αυτά είναι, μας ανησυχούν βαθύτατα. Οπότε μπορείτε να υπολογίζετε σε εμά για την τελειοποίηση του καταλόγου των προϋποθέσεων της αρεσιμότητας, αλλά θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν θέλουμε εσφαλμένες πολιτικές κρίσεις για το κατά πόσο συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Γι' αυτό ίσως μια εκτελεστική πράξη είναι προτιμότερη από μια καταξουσιοδότηση πράξη, όταν ιδιαίτερα υπάρχουν κάποια πολιτικά θέματα. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει να διευκριστεί περαιτέρω στο νομοθετικό κείμενο για το θέμα των συμβολών, των συνεισφορών με βάση το, για το βασικό κίνδυνο και να προσέξουμε ιδιαίτερα την ε, έκθεση σε δημόσιο χρέος. Επίσης, ε, είπε ότι θα πρέπει να είναι προκυκλικές οι συνεισφορές. Νομίζω ότι όμως οι εξπόσεις συνεισφορές θα μπορούσαν να, να ε, ρυθμιστούν ώστε να βγάλουμε το προκυκλικό ζήτημα. Επίσης, ε, είπες να αξιολογήσουμε την καταλληλότητα του στόχου 0,8% σε τακτική βάση. Επίσης, ε, λέμε να δώσουμε στο ΕΝΤΙΣ και στο Ταμείο ε, μια τραπεζική άδεια, να προσθέσουμε ένα backstop αντίστοιχο με αυτό που ισχύει για, για το SRM, ώστε να έχουμε υψηλή εμπιστοσύνη σε όλες τις χώρες, δηλαδή ένα ευρώ στην α χώρα να ισχύει το ίδιο με ένα ευρώ σε άλλη χώρα, όποια και είναι η χώρα αυτή. Να είναι ίδιος ο βαθμός προστασίας και ασφάλειας. Τώρα αυτός ο κοινό ε, μηχανισμός ασφαλείας θα μπορούσε να ε, εισαχθεί σταδιακά ανάλογα με το βαθμό αμοιβαιοποίησης της προστασίας των καταθετών και να δούμε πώς θα ε, καταμετρούμε και θα παρακολουθούμε τους κινδύνους, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα συστημικά ιδρύματα, να λάβουμε υπόψη το θέμα των τραπεζών του Big to Fail, Deutsche Bank και άλλες. Και επίσης να, να καλυφθεί το θέμα του συσχετισμού των συστημάτων. Ω προ το χρονικό το χρονισμό, το χρονοδιάγραμμα, προτιμούμε να παρατεθεί η προθεσμία για τις τροπολογίε. αλλά πριν από αυτό θα πρέπει να συναντηθούμε με τους συντάκτες τη μελέτη επιπτώσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να έχουμε μια κοινή ερμηνεία και να αντιληφθούμε όλα τα επιμέρου στοιχεία τη μελέτη αντικτύπου. Όπω θα καταλάβατε, θέλουμε να συμμετέχουμε σε μια συμμαχία όσων επιθυμούν πραγματική πρόοδο για το θέμα αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη. Και πολύ συμμερίζω αυτό το πνεύμα. Να δημιουργήσουμε λοιπόν αυτή τη, τη συμμαχία των προθήμων και να μην υποχωρούμε σε αυτούς που θέλουν να τορπιλήσουν αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε Μαρκο Ναι, ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση που παρουσιάζει που φαντάζομαι χρειάστηκε εβδομάδες και μήνες για να ολοκληρώσει. Έγιναν ε, πολλές συναντήσεις, ενημερωθήκαμε για τις διάφορες δυνατότητες, διαβάσαμε την πρόταση της Κομισιόν και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση γιατί το βασικό πρόβλημα αυτή της νομοθεσία ουσιαστικά είναι το βασικό πρόβλημα της πρόοδου της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η έλλειψη πολιτικής συμφωνίας, ε, διαφορετικά πολιτικά οράματα, διαφορετικά μοντέλα ε, μεταξύ των διαφορών πολιτικών δυνάμεων. Αυτές οι διαφορές κατέστησαν ορατές και θα, θα στον οράτε και στο πλαίσιο αυτή τη έκθεση ε, που αφορά την ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση, ένα από τα σημαντικότερα έργα εντό Ευρωζώνη, για το οποίο ε, έχουν επενδύσει πολλοί οι κυβερνώντε. Ένα από τα έργα τα οποία θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο να σταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα, να το καταστήσει πιο ασφαλές. Πιστεύω ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος που θα έχουμε στο νου μας, ε, ε, εξετάζοντας το κείμενο αυτό. Προσωπικά σε γενικές γραμμές ε, θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο παρότι η προσέγγιση της δικής μου ομάδας και εμού ως ε, ε, σκιώδης συγκεκριτή θα είναι θετική, θα ασκήσουμε επικοδομητική κριτική και πολύ συγκεκριμένη και ακριβή. Ωστόσο δεν βλέπω να υπάρχει δυνατότητα πολιτικής συμφωνίας είτε στο Κοινοβούλιο είτε στο Συμβούλιο όταν μιλάμε για ένα τέτοιο νομοθέτημα το οποίο θα μπορούσε να σταθεροποιήσει πραγματικά και να βελτιώσει το σύστημα. Ο φόβος είναι ότι για άλλη μια φορά ε, αυτή η οροσυρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα δημιουργήσει κάτι μικρό το οποίο θα υπονομεύσει τη σταθερότητα. Θα μας δώσει να δούμε δηλαδή ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία διαφωνίας ε, τα οποία αποτελούν τα τροτά μας σημεία. Όσον αφορά την πρότασή σας, για την οποία θα κάνουμε εμεί αντιπροτάσει μέσω τροπολογιών, πρόκειται για μια βάση εργασιασμένη, αλλά κατά την άποψή μου θα υπο, υποβαθμίσει την ίδια δύναμη πρόταση δομή ε, τη πρόταση τη Κομισιόν. Ε, κάποιες βελτιώσεις θα ήταν ε, να, μειωθούν οι τρει σε δύο φάσει για το όλο έργο. Αυτό είναι μια ε, καλή πτυχή απλούστευση ώστε να επιτευχθούν τα αποτελέσματα γρήγορα, να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο να λειτουργεί δηλαδή πλήρω, Ωστόσο, από την άλλη πλευρά διακρίνω και όσον αφορά τη χρήση της ορολογίας ε, και στις τροπολογίες ε, βλέπω ότι υπάρχει κίνδυνος να καταπνίξουμε την πρόταση αυτή. Ε, όταν εσείς μιλάτε για liquidity support ε, αντί για funding, όταν αντικαθιστέτε τον όρο excess loss cover όταν ε, εξέλιφεται όλες τις αναφορές ε, στην fully mutualized approach εκεί βλέπω εγώ διακρίνω ένα κίνδυνο ε, να καταπνίχει η πρόταση. Για πολύ συγκεκριμένα θέματα τώρα, πέραν της δομής, η οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκη και συνεπώς αναποτελεσματική, αυτό το σύστημα του DIF που υποδιαιρείται σε υποταμεία μεταξύ των διαφορών συστημάτων και των εθνικών ταμείων είναι πολύ περίπλοκο για να είναι αξιόπιστο, για να είναι πιστευτό κατά την απόψή μου. Πράγματι αυτό που διαβάζω στην πρόταση είναι σωστό. Η joint capacity, δηλαδή η αμοιβεοποιημένη δυνατότητα θα αντιστοιχεί μόνο στο 0,2% του συνόλου των καταθέσεων που θα πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο εγγύηση εντό του συστήματο. Φαίνεται λίγο όταν μιλάμε για ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει σε περίπτωση συστημικής κρίσης. Και ακόμη και να αυξήσουμε το ποσοστό, θεωρώ το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Ακόμα και αν η joint capacity φτάσει στο 0,8% των καταθέσεων. Γιατί, διότι λείπει ένα θεμελιώδη σημείο κατά την απόψή μου για να γίνει πιστευτή αυτή η πρόταση. Ε, ένας ε, δημόσιος μηχανισμός ασφαλείας. Ε, το ξανασυζητήσαμε και παλιότερα, αυτό το backstop ε, συναντηθήκαμε με κάποιον εκπρόσωπο των ΗΠΑ που απάντησε στο ερώτημά μας κατά πόσο είναι σημαντικό να υπάρχει ένα public backstop το οποίο να καθιστά αξιόπιστο το γεγονός ότι σε περίπτωση συστημικής κρίσης το εργαλείο αυτό πράγματι θα χρησιμεύσει, θα είναι λειτουργικό και σε κάθε περίπτωση οι ε, τρεχόμενοι λογαριασμοί των πολιτών ε, δεν θα διατρέχουν κίνδυνο, θα είναι ασφαλείς. Η τραπεζική κρίση στις ΗΠΑ το 2008 κόστησε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ στους Αμερι... Ε, δολάρια στους Αμερικανούς το να θεωρούμε ότι θα μπορούμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα συστημικής κρίσης χωρίς public backstop, κατά την άποψή μου, είναι τρέλα. Είναι κάτι που δεν είναι πιστευτό. Έχουμε ένα θεσμό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εντός Ευρωζώνης, που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να λειτουργεί ως public backstop έσχα της λύσης στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Μόνο κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δώσει αξιοπιστία στο εργαλείο αυτό και να καταστήσει πραγματικά τους τροχούμενους λογαριασμούς των πολιτών ασφαλείς. Θα μπορούσε να αποτελέσει απάντηση πιστική όσον αφορά τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης και θα μπορέσει πραγματικά να ολοκληρώσει την Τραπεζική Ένωση. Χωρίς τέτοια προσέγγιση, χωρίς τέτοιου είδους εργαλείο, ε, το οποίο μπορεί να κάνει μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι ο μόνος οργανισμός που μπορεί να τυπώσει ευρώ και μπορεί να πει, ξέρετε, με τα νούμερα αυτά που βλέπετε στους τρεχόμενους λογαριασμούς σας ε, εγγυώνται από εμάς που τυπώνουμε χαρτονομίσματα. Είναι ο μόνος δρόμος, η μόνη οδός ε, για να λειτουργήσει σωστά το εργαλείο αυτό. Τώρα, όσον αφορά την εισαγωγή των payment commitments, και εδώ θέλει ένα ερωτηματικό. Είμαστε βέβαιοι ότι σε περίπτωση συστημικής κρίσης τα συστήματα θα είναι σε θέση, οι θα είναι σε θέση να ε, τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις πληρωμών, τα payment commitments. Έχω ένα ερωτηματικό γι' αυτό. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία, τα οποία θα ήθελα να αναλύσουμε και τα οποία ήθελα να τονίσω. Εμείς ως ομάδα θα θέλαμε να συνεργαστούμε για να βελτιωθεί αυτή η πρόταση η οποία πιστεύω στην παρούσα εμβριακή φάση δεν είναι επαρκής για να διασφαλίσει τη σταθερότητα, ούτε για να διασφαλίσει τα όσα χρειαζόμαστε για να βελτιώσουμε και να σταθεροποιήσουμε περισσότερο το σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω τον ομιλητή του ΙΕΝΕΦ, οπότε να ξεκινήσουμε με το ΚΑΤΣΔΙΑ. Οι πρώτος ομιλητής, ε, Μπολχερ Μπάλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την Εστέρ Ντελάγκη για τη δουλειά που έκανε. Βεβαίω το Συμβούλιο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τις ε, διαβουλεύσεις. Ε, Εν τω μεταξύ η εισηγήτρια νομίζω πως ε, τόλμησε θα έλεγα. Πρόκειται για μια καλή αφετηρία για την περαιτέρω συζήτηση και ως τέτοια πρέπει να την δούμε. Η κυρία Ντελάνκη εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο ακριβώς για να δει τα ευαίσθητα εκείνα σημεία στα οποία χρειαζόμαστε αποτελεσματικές λύσεις. Αυτά είναι, κατά την άποψή μου, η αναγνώριση της λειτουργικότητας των εθνικών συστημάτων ασφάλισης καταθέσεων, τα οποία μπορούμε ακόμα να εκμεταλλευτούμε και μετά βεβαίως ο περιορισμός του ηθικού κινδύνου και κατόπιν η ανάγκη να μειωθεί ο κίνδυνος πριν οι φυστάμινοι κίνδυνοι μεταφερθούν σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο και βεβαίως μια καλύτερη κατανόηση των περαιτέρω ε, των, βημά, των συνεπειών των περαιτέρω βημάτων προς μια ευρωπαϊκή εναρμόνιση. Σε γενικές γραμμές λοιπόν Πρόκειται για σημεία τα οποία είναι όλα εξαιρετικά πολιτικά και θα πρέπει νομίζω να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στην συζήτησή τους. Ε, τα ανοιχτά σημεία του Ήλις ε, νομίζω δεν έχουν απαντηθεί επαρκώς από την ε, ανάλυση της Κομισιόν η οποία δεν είναι αξιολόγηση αντικτύπου και αφήνει αναπάντητα ερωτήματα όπως η επίδραση στους ίσους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, η αποτίμηση των υφισταμένων κινδύνων και τα διάφορα εθνικά συστήματα που υπάρχουν ήδη. Νομίζω λοιπόν πως έχουμε μία στέρη βάση εδώ πέρα. Η συγγήτρια πράγματι πηγαίνει από μια επιλογή αντασφάλισης σε μια επιλογή ασφάλισης. Ε, εμείς υποστηρίζουμε την εισηγήτρια και την προσέγγιση της ε, να αποστείλουμε και ένα μήνυμα και στις άλλες επιτροπές για να αναζητήσουμε μια ισορροπημένη λύση. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπερές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια που κατέθεσε μια πρόταση πολύ σημαντική για να γίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαντικός παράγος στην όλη συζήτηση. Να συμμετέχουμε ενεργά στην όλη συζήτηση και να διαμορφώσουμε μια θέση που θα αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω συζήτηση. Λυπούμε πάντως που η πρόταση αυτή που την περιμέναμε πώς και πώς διέρευσε και σε κάποιους δημοσιογράφους και μάλιστα πριν την λάβουν προς μελέτη οι ευρωβουλευτές, κάτι που δημιουργεί κάποιο πρόβλημα λειτουργίας. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το πρόβλημα το βασικό. Το βασικό ζήτημα είναι ότι η προσέγγιση που μας προτείνει η συγγήτρια είναι από τη βάση προς τα πάνω, από κάτω προς τα πάνω, ενώ η Τραπεζική Ένωση υιοθετούσε μια διαφορετική προσέγγιση, αντίστροφη, από πάνω προς τα κάτω. Όταν θεσπίσαμε το μηχανισμό της Τραπεζικής Ένωσης είχαμε μια συνολική προσέγγιση, συστημική σχεδόν, για το ποιοι θα πρέπει να είναι οι τρεις πυλώνες μιας Τραπεζικής Ένωσης. Ε, είδαμε ότι για τον τρίτο πυλώνα της εγγύης καταθέσεων υπήρχαν ανησυχίε ε, σε πολλές χώρες. Και είχαμε την αίσθηση ότι ε, ξεκινήσαμε αυτές τις ανησυχίες κάποιων χωρών ε, για να βρούμε λύση. Και θεωρώ ότι σε αυτή την πορεία υπάρχει ο κίνδυνος, οι ίδιοι στόχοι της Τραπεζικής Ένωσης να παραμεριστούν. Δηλαδή έχουμε ένα σύστημα που ίσως ε, περάσει, αλλά ίσως χάσει τον τελικό του στόχο, που είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ασφάλεια που μπορεί να τους προσφέρει το σύστημα και που αναγκαστικά εδράζεται σε μια γνήσια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεν θα επισέλθω τώρα σε λεπτομέρειες για την αρεσιμότητα. Θα έχουμε την ευκαιρία με τις τροπολογίες μας να τελειοποιήσουμε αυτό το σημείο και χαίρομαι για την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Καταρχήν, ανησυχώ για την τρίτη φάση της πλήρους αμοιβαιοποίησης που την αφήσαμε κατά μέρος ή την αφήσαμε στην κατεξουδότηση πράξης. Ήθελα να συμπεριληφθεί εγώ από την αρχή στο, στο συνολικό σχεδιασμό, ώστε να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Και επίσης ενώ εμείς έχουμε αυτή τη συζήτηση, το Συμβούλιο φαίνεται ότι έχει κολλήσει στο θέμα του backstop, του μηχανισμού ασφαλείας. Βέβαια, θα παρακολουθούμε εκ του και στα θέματα, αλλά χαίρομαι που επιτέλους ε, μπήκαμε στο ψαχνό της συζήτησης, στο βασικό της πυρήνα και στα σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ κυρία Μπέρες. Ο Πέτερ Σάιμον έχει το λόγο τώρα, ο αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν ξεκίνησε εδώ η συζήτηση για το ΕΔΙΣ, εγώ στον πρώτο γύρο των συζητήσεών μας είχα πει πως στόχος μας πρέπει να είναι να έχουμε περισσότερη σταθερότητα σε όλες τις χώρες. Αυτό σημαίνει πως δεν βοηθάει κανέναν να έχουμε ένα υψηλότερο γενικό επίπεδο σταθερότητας, αλλά στις μεμονωμένες χώρες να έχουμε χαμηλότερο επίπεδο σταθερότητας. Αυτό προσπάθησε να το λάβει υπόψη η κυρία Ντελάγκε με, κάνοντας έναν διαχωρισμό. Έναν διαχωρισμό αφενός ο οποίος ε, δίνει την δυνατότητα αφενός να συνεχίσουν να υπάρχουν και στο μέλλον τα σταθερά εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων. Ταυτόχρονα να υπάρχει και αλληλεγγύη, κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνος στο Κοινοβούλιο. Η ομάδα μας, οι περισσότερες ομάδες εδώ πέρα αναγνωρίζουν ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και περισσότερη ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά στη διαμόρφωση μετά πρέπει να δούμε κάποια πράγματα πιο λεπτομερώς και εδώ πέρα θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για την περαιτέρω συζήτηση και να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Εάν στο σύστημα αυτό καταλήξουμε στο αποτέλεσμα ότι υπάρχει πρόβλημα σε μια χώρα που χρειάζεται ευρωπαϊκή ενίσχυση και άρα μιλάμε για τον ευρωπαϊκό κορβανά που θα πρέπει να πληρώσει, θα πρέπει να δούμε πώς θα ξαναγεμίσει αυτός ο κορβανάς γρήγορα. Γιατί μπορεί βεβαίως και πιθανότερο είναι να ακολουθήσει αμέσως άλλη μια κρίση. Οπότε θα πρέπει να έχει ένα preferred creditor status, ε, όπως και το IMF, e για να διασφαλίσουμε ότι το συντομότερο δυνατόν θα είναι επαρκή τα κονδύλια. Δεύτερη ερώτηση που προκύπτει, αν δούμε ακριβώ αυτόν τον κόρβανα, έχουμε την δεύτερη πτυχή, τα εθνικά ευρωποιημένα πλέον τι γίνεται στις χώρες οι οποίες έχουν ήδη τέτοια εθνικά συστήματα. Έχουν περισσότερες εγγύησεις ή μόνο τα μία εγγύησεων ή μόνο ένα. Υπάρχουν επιχειρήματα και για τα δύο. Μία τρίτη ε, παρατήρηση αφορά το θέμα του για ποιο σκοπό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα λεφτά και να ευχαριστήσω την Έστερ που είπε πως θα πρέπει να υπάρχουν οι δυνατότητες και για εναλλακτικά μέτρα. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και εκτός ε, των ε, συστημάτων ε, διασφάλισης, δηλαδή εναλλακτικά μέτρα σε άλλες χώρες και για άλλες τράπεζες που θα πρέπει να είναι δυνατά. Επίσης θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό να σκεφτούμε την δυνατότητα η εγγύηση των ε, καταθέσεων να χρησιμοποιηθεί εάν σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας τράπεζας ολόκληρη ε, λογαριασμοί, σχέσεις με πελάτες μεταφέρονται από την μία τράπεζα στην άλλη και τότε υπάρχει κάποιο κόστος και θα πρέπει να προστατεύεται ο, πελάτης ε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και νομίζω θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και για αυτόν τον σκοπό την ε, ασφάλεια των ε, καταθέσεων για να έχουμε ακόμη καλύτερη προστασία του πελάτη, του καταθέτη, από το ότι αν ήταν εξαρτημένος από μία μόνο τράπεζα. Τέλος, είπα όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι υπάρχει αυτή η πρόταση για να παραταθεί η προθεσμία. Αναμένω τη συζήτηση λοιπόν με την εισηγήτρια. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος τώρα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια πρώτα απ' όλα, της οποίας η έκθεση εμένα με εξέπληξε, εξέπληξε θετικά γιατί περιέχει διάφορες σημαντικές πτυχές για την συζήτηση και έχουμε ένα δύσκολο θέμα το οποίο μπορεί να λάβει τώρα νέα όθηση. Εγώ ζήτησα τον λόγο γιατί ο συνάδελφος Φίλιπ Λάμπερτς ε, δυστυχώς δεν είναι πια στην ε, έθεσε ρητός ε, το θέμα προς τους Γερμανούς συναδέλφους. Νομίζω πως εδώ στο παρελθόν Καλά κάναμε ότι αντιμετωπίζαμε δηλαδή τα προβλήματα ευρωπαϊκά σε μια ευρωπαϊκή διάσταση και όχι με ε, εθνικά ε, γυαλιά. Τώρα βλέπω είναι πάλι εκεί ο συνάδελφος. Λοιπόν, αν υπάρχουν κίνδυνοι και πράγματι υπάρχουν σε όλες τις χώρες ε, κίνδυνοι, πράγματι είναι να αναφέρονται, αλλά νομίζω πως η αρχή και το πνεύμα είναι το εάν το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το κατάλληλο επίπεδο για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και ποιο είναι το κατάλληλο μέσο. Έχουμε στις ευρωπαϊκές συνθήκες ε, την αρχή της επικουρικότητας ε, και βεβαίως ε, το να λέμε έτσι ότι έχουμε βρει μία λύση η οποία είναι η κοινοτικοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων ε, και ως διαμαγεία θα λυθούν όλα δεν είναι τόσο αυτόματο. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι σωστές απαντήσεις για να δούμε ε, για να αντιμετωπίσουμε τους υφιστάμενους ε, κινδύνους. Και θα ήθελα να πω πως οι προτάσεις εδώ πέρα που έχει βάλει σε αυτό το πακέτο η Εστέρ πηγαίνουν προς την σωστή κατεύθυνση με ξεκάθαρα κριτήρια Έχουμε κάποια χαρακτηριστικά, παραδείγματος χάρη, οι ειδικοί λένε εδώ και χρόνια το ότι τα κρατικά ομόλογα εδώ και χρόνια έχουν ένα θέμα με τα ίδια ε, κεφάλαια, κάτι το οποίο λειτουργεί, δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά και θα πρέπει να καταφέρουμε νομίζω να βάλουμε όλες αυτές τις πτυχές σε ένα πακέτο και έχουμε νομίζω μια νέα βάση για συζητήσεις ε, και θα ήθελα να απευθύνω έκκληση όπως σας είπα να μην βλέπουμε τα πάντα με εθνικά ε, γυαλιά ο καθένας αλλά με μια ευρωπαϊκή οπτική για να λάβουμε υπόψη επίσης και το θέμα της αναλογικότητας που πρέπει να παίξει ένα ρόλο δηλαδή τα μέτρα πρέπει να είναι και αναλογικά με το πρόβλημα να λάβουμε υπόψη βεβαίως και τις υφιστάμενες τις υπάρχουσες ε, δομές ε, που ήδη λειτουργούν ε, τα εθνικά δηλαδή συστήματα ασφάλισης καταθέσεων τα οποία δεν πρέπει να καταστραφούν αυτό θα ήταν λάθος ακριβώς το θέμα είναι και όπου δεν υπάρχουν τέτοια συστήματα εγγύησης καταθέσεων να δημιουργηθούν έτσι ώστε όλοι οι καταθέτες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι διασφαλισμένοι. Indeed. Σας ευχαριστώ, κύριε Τόιρερ. Δεν βλέπω άλλο συνάδελφο να θέλει το λόγο, οπότε να ξαναδώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Ντελάνκε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που υπογράμμισαν ακριβώ τι ευαισθησίε που υπάρχουν για το θέμα αυτό. Πάντως χαίρομαι και εκτιμώ ιδιαίτερο την ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση που είχαμε μεταξύ μας. Και Ευχαριστώ και του συναδέλφου που έκαναν πολύ τεχνικέ παρατηρήσει, ουσιαστικέ επί του περιεχομένου, γιατί θα μα βοηθήσουν να προχωρήσουμε. Τεχνικά θέματα, όπω το book transfer ως εργαλείο στα χέρια τη SRB, αλλά σε συνεργασία φυσικά με τα εθνικά συστήματα, δεν ξέρω πώ αλλιώ θα μπορούσαμε να το κάνουμε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, γιατί τέτοιου είδου ε, προτάσει πραγματικά εμπλουτίζουν την έκθεση. Και σα ευχαριστώ. Ε, να κάνω κάποια σχόλια για τα, τους φίλους μας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έκαναν καλά τη δουλειά τους και μάλιστα κατάφεραν να εξασφαλίσουν ε, κάποιες, ε, κάποια σχέδια της έκθεσης, αλλά με πρόσβαλε το σχόλιο της συντονίστρια των σοσιαλιστών που φαίνεται ότι κατηγορείται η συγκεκριμένη Μα εδώ διαρροέ έχουμε προ όλε κατευθύνσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν φταίω εγώ που έγιναν αυτέ οι διαρροέ προ δημοσιογράφου. Και άλλωστε ήταν παλιέ οι διαρροέ. Ήταν τα πρωταρχικά πρωτόλιες προτάσεις γιατί βλέπετε ότι στη διαρροή που έγινε του δημοσιογράφους είχαμε διαφορετική διατύπωση, πολύ πιο αυστηρή από τη διατύπωση που τελικά διάλεξα στην οριστική μου έκθεση που σας μοίρασα. Και μάλιστα εγώ την οριστική μου έκθεση μόλις τώρα την ε, ολοκλήρωσα και σας διαβεβαιώ ότι δεν, έκανα, δεν είμαι εγώ η υπεύθυνη για τις διαρροές. Και δεν ξέρω από πού προήλθαν οι διαρροές, πάντως σας διαβεβαιώ κύριε στους σοσιαλιστές ότι αλλού έπρεπε να σηκώσετε το δάχτυλο και να δείξετε προς άλλη κατεύθυνση για τις διαρροές. Τώρα για το περιεχόμενο της έκθεσης, πολύ ευχαρίστως να επανεξετάσουμε την ερμηνεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη μελέτη επιπτώσεων που έκανε. Οπότε θα βρούμε κάποιο χρόνο και τρόπο για να συνεννοηθούμε με τους κοιόδους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως είναι σαφές ότι στη σελίδα 4 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η υποχρεωτική αντασφάλιση ε, ξεπερνά το, το υποχρεωτικό σύστημα και μιλάει για κοντά στα αμοιβεοποιημένα κεφάλαια. Δεν είναι δικά μου αυτά τα λόγια, είναι λόγια της ε, μελέτης αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της συμπληρωματικής αξιολόγησης που έκανε μάλιστα. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί η πρόθεσή μου και η φιλοδοξία μου που δεν, ε, που δεν, ήταν να κάνω αυτό το εργαλείο ε, μικρότερο ή επουσιώδες. Θα πρέπει να έχει την ίδια ισχύ. Ε, δεν θα δεν θα ήθελα την καραμπίνα να την κάνω πιστολάκι, αλλά ούτε θα είναι και μπαζούκα που θα λύσει όλα τα προβλήματα έλλειψη αξιοπιστία ή ε, σταθερότητα που έχει ο τραπεζικό κλάδο. Αλλά συμφωνώ μαζί σου ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση. Αλλά όσο ό,τι αφορά τι αναλογίε, θα πρέπει να είμαστε σαφεί. Η παρατήρηση του Φίλιπ Λάμπερτ που είπε τι γίνεται για τις ε, πιο συστημικές μεγάλες τράπεζες και πόσο κατάλληλη είναι η δεύτερη φάση που προβλέπεται για αυτές τις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Ας είμαστε ρεαλιστές, αυτές ε, οι μεγάλες ε, τράπεζες θα πάνε στο μηχανισμό εξυγίανσης και όχι στο μηχανισμό αφαιρεγκαιότητας. Αυτά θα τα πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας. Επίσης, το θέμα του χρονοδιαγράμματος και της παράτασης ε, της προθεσμής και της τροπολογίας χαίρομαι που διευκρινίστηκε και διευθετήθηκε. Είμαι κι εγώ ελαστική. Η φιλοδοξία του προτινόμενου συστήματος από μένα δεν είναι χαμηλότερη από τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. συζητήσαμε την ισχύ του. Δεν συρρυκνώνω ε, την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ δεν αγγίζω το 0,8%. Το 0,4% των εθνικών DGS και το 0,4% του Ευρωπαϊκού Ταμείου καταλήγουν στο ίδιο πράγμα. Είναι αλληλένδετα ε, και συνεργάζονται στενά με το ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα. Και αυτό που είπατε κύριε Παπαδημούλη, παρα, το 0,4 του Ευρωπαϊκού Ταμείου, ε, δεν ε, αφορά το 0,4 του Εθνικού Ταμείου. Και αν είχαμε κάτι τέτοιο θα είχαμε περικοπή τη ισχύω του συστήματος, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι έτσι εγώ την νομοθεσία. Εγώ δεν άγγιξα καθόλου, δεν μείωσα καθόλου το 0,8 της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ισχύ του συστήματος. Εγώ ήθελα να βρούμε έναν τρόπο για να οργανώσουμε τις ευθύνε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι ο μόνο τρόπος που θα ε, λειτουργήσει το σύστημα. Μερικοί μπορεί να αποκαλούν αυτό το θέμα ηθικό κίνδυνο, άλλοι να μην προτιμούν αυτή τη διατύπωση. Πάντω θα πρέπει να βρούμε τρόπο ώστε το σύστημά μα να στηρίζεται στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την ευρωπαϊκή ευθύνη, αλλά και στην εθνική ευθύνη. Και αυτή είναι η απάντησή μου και προ του σοσιαλιστέ. Όταν αναφερθήκατε στο εθνικό επίπεδο, 100% του προβλήματος που βλέπουμε στο σύστημα θα επιληθεί. Και αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα οργανώσουμε και θα καταμερίσουμε τις ευθύνες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό ενιαίο σύστημα που θα έχει την ίδια ισχύ και εμβέλεια με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σιλβί, το πλαίσιο της αφαιρεγγιότητας είναι κάπως δύσκολο, ακαθόδες και το να τα αφήνουμε στα χέρια των Υπουργών Οικονομικών είναι ούτως ήδη δύσκολο το θέμα. Πολλό δε μάλλον να το αφήσουμε στα χέρια των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, ακόμη χειρότερο. Πάντως ε, συμφωνώ ότι όλοι οι εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι η αφαιρεγκαιότητα είναι κλειδί για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και σίγουρα ο κατάλογος αρισιμότητας δεν θα πρέπει να γίνει πρόσχημα ε, για την απραξία. Θέλουμε ένα κατάλογο προϋποθέσεων που να είναι κατάλληλος για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύσεων. Και σίγουρα η αφαιρεγγιότητα ανήκει σε αυτά τα κριτήρια. Και το ατού της πρότασης είναι ότι σε ό,τι αφορά τη μείωση του κινδύνου, γιατί με ρώτησε Σιλβία θα είναι παράλληλο το σύστημα ή θα είναι ένα σκληρό όριο ή ένας, ένα τέρμα στο σύστημα. Το θέμα είναι να έχουμε μία φάση πλήρους στήριξης ε, της ρευστότητα. Και να το δούμε αυτό και χρονικά. Επίσης, τέθηκε μία ερώτηση από τον κύριο Ζάιμον. Ε, έφυγε βέβαια στο μεταξύ και θα του το διευκρινίσω διμερός. Και τέλος, γιατί τη σειρά ικανοποίηση ε, ε, στην περίπτωση διαδικασίας αφαιρεγκιότητας και αν θα είναι αντίστροφη από ότι η εκταμίευση από το Ταμείο. Πάντως, ε, περιμένω συνέχιση των συζητήσεων, αλλά σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Δεν είναι το τέλος σίγουρα, είναι μόνο η αρχή, παρόλο που η διαδικασία ήταν ήδη αρκετά χρονοβόρα. Ευχαριστώ κύριε Λάγκη, συμφωνώ απόλυτα ότι όντω. Ε, αυτή είναι μόνο η αρχή. Γιατί... την Κομισιόν αν θέλει να μιλήσει. Σύμφωνα με τη γραμματεία, ε, συμφωνήσαμε να μην δώσουμε τον λόγο μέχρι στιγμή στην Κομισιόν, εκτό αν πραγματικά ενδιαφέρεται να παρέμβει. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πριν σας δώσω την προθεσμία για την εκθεσία αυτή, να πούμε κάτι για την προθεσμία της Τραπεζικής Ένωσης, ε, η προθεσμία τροπολογιών για την Τραπεζική Ένωση θα είναι 16 Δεκεμβρίου. Εξέταση των τροπολογιών στις 12 Ιανουαρίου, ψηφοφορία 25 Ιανουαρίου στην Επιτροπή και ψηφοφορία στην Ολομέλεια στις, στην δεύτερη Ολομέλεια του Μαρτίου. Όσον αφορά για 16 ε, Δεκεμβρίου για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων, υποβολή τροπολογιών 16 Δεκεμβρίου, 25 Ιανουαρίου εξέταση των τροπολογιών και δεν έχει ακόμα οριστεί η ψηφοφορία στην Επιτροπή. Και τέλος, ανακοινώνω ότι σε μισή ώρα θα γίνει μια ανοιχτή ε, συνεδρίαση συντονιστών που θα λάβει χώρα σε αυτήν εδώ την αίθουσα στις 12 και 4 σε μισή ώρα. Οπότε διακόπτουμε για μισή ώρα. Ευχαριστώ πολύ.